So, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε έτσι ώστε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Πρέπει να δεχτούμε τις ε, προτάσεις των εισηγητών, συγγνώμη, των συντονιστών από τη χθεσινή του συνεδρίαση. Και μετά θα περάσουμε στα 17 και 18 και θα συζητήσουμε λοιπόν από κοινού τις δύο εκθέσεις. 17 και 18. Πρώτο ζήτημα. Θα υπάρξει μία έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο την 10η Ιουνίου, ούτως ώστε να εγκρίνουμε το πακέτο για το άσυλο. Διότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ψηφίσει για το θέμα αυτό τον Ιούνιο και επομένως εμείς οφείλουμε να κάνουμε την 10η Ιουνίου ε, στο Στρασβούργο μια έκτακτη συνεδρίαση. Οι συντονιστές αποφάσισαν να ζητήσουν έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας με θέμα ε, των ε, πίνακα επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα της δικαιοσύνης σε όλες τις χώρες μέλη. Επίσης, συμφώνησαν οι συντονιστές να καλέσουν την νομική υπηρεσία για δήλωση ενώπιον της Επιτροπής μας την 6η Μαΐου σχετικά με την ε, έκθεση Μακοβέη για τις κατασχέσεις και να συζητήσει το θέμα ε, της έκθεσης την 7η Μαΐου στην Επιτροπή μας. Επίσης, ε, αντιπροσωπεία θα μεταβεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο ε, Εξάρτησης από Ουσίες. Επίσης, προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, ακολουθούμενη από ψήφισμα σχετικά με την εφαρμογή της εσωτερικής στρατηγικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερη έκθεση, επί μάλλον της δεύτερης έκθεσης της Επιτροπής. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν συμφωνείτε με τις συστάσεις των συντονιστών. Δεν βλέπω κάποιον να έχει σχόλια, επομένως ε, θεωρούνται αποδεκτές οι συστάσεις αυτές και επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε άμεσα με την εξέταση των σημείων 17 και 18. Κοινή συζήτηση για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς επίσης και τη χρηματοδότηση της θερμοκρατίας, έκθεση Σαρτζεντίνη. Και το άλλο θέμα, πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών με εισηγητή τον κύριο Κίρκχοπ. Η Κομισιόν έχει υποβάλει ήδη τις ε, προτάσεις της στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίηση χρηματοδοτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων, ε, καθώς επίσης και τον κανονισμό για τις πληροφορίες που συνοδεύουν τι μεταφορέ ε, χρηματικών ποσών και οι δύο προτάσεις αφορούν την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων και της τρομοκρατίας μέσω της καταπολέμησης ε, του ξεπλήματος ε, χρήματος. Οι δύο προτάσεις ε, στην ουσία αναφέρονται στην έννοια και την αντίληψη που έχουμε όσον αφορά το φορολογικό έγκλημα κλπ. κλπ θα αφήσω στους ε, εισηγητές ε, ε, να αναφερθούν στο θέμα αυτό. Όμως πρέπει να σας πω ότι έχουμε λάβει επιστολή από την Επιτροπή Μελέτης του άρθρου 29, από τον πρόεδρο της Επιτροπής, και πρέπει να σας πληροφορήσω επίσης ε, ότι η Επιτροπή ΕΚΟΝ ε, έχει αμφισβητήσει την, ε, δικαιο... την αρμοδιότητα της ΛΥΜΠΕ για τα δύο αυτά θέματα. Θα συζητηθούν αυτά στη διάσκεψη των Προέδρων. Θα δώσω πρώτα τον λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής για μια παρουσίαση των δύο θεμάτων και μετά στους εισηγητές και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιον εκπρόσωπο έχουμε. Φόν και Μακ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Oh, better. Okay. Excuse. Τώρα με ακούτε, ε? Ωραία. Θα είμαι σύντομος, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Αλλά ευχαρίστως να απαντήσω σε ερωτήσεις ε, που ίσως γίνουν. Θα ήθελα να τονίσω τα βασικά ζητήματα που υπάρχουν στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας. Πρώτο σημαντικό πράγμα που πρέπει να πούμε είναι πως έχουμε αναθεώρηση φυστάμενης οδηγίας, οπότε δεν είναι κάτι το καινούριο. Έχουμε εξελίξει πράγματα τα οποία υπήρχαν ήδη, αλλά δεν πρόκειται περί επανάστασης ούτε περί ενός εντελώς νέου μέσου. Κάναμε λοιπόν αυτή την αναθεώρηση για δύο λόγους ουσιαστικά. Ο πρώτος είναι πως πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθούμε τη διεθνή πρότυπα της ε, Διεθνούς ε, Ομάδας Δράσης για την ε, χρηματοπιστωτική δράση και ακριβώς αυτή η ομάδα αναθεώρησε τα πρότυπά της και θεωρήσαμε σωστό να κάνουμε και εμείς το ίδιο και κάναμε και τη δική μας αξιολόγηση της λειτουργίας της τρίτης οδηγίας πολέμησης του ξεπλήματος χρήματος και είδαμε κάποια ζητήματα που άξιζε να βελτιωθούν με βάση, όπως είπα, τη δική μας αναθεώρηση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα άλλων αυτών. Υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί τομείς όπου έγιναν αλλαγές και θα επικεντρωθώ σε αυτούς και ξεκινάμε βεβαίω με ζητήματα πεδίου εφαρμογής το οποίο έχουμε διευρύνει στην τέταρτη οδηγία για, το ξέπλυμα χρήματος έχουμε συμπεριλάβει όλες τις μορφές τζόγου και ο στόχος, ο λόγος είναι πως ε, σε πολλά κρατημέλη ήδη συμβαίνει αυτό υπάρχουν ενδείξεις πως υπάρχουν κίνδυνοι ξεπλήματος χρήματος που σχετίζονται με κάποιες μορφές τζόγου που δεν ε, καλύπτονταν, ε, γιατί μέχρι στιγμής καλύπτουμε καζίνος στο ίντερνετ και στον πραγματικό κόσμο, αλλά τα υπόλοιπα όπως το στοίχημα της χάρη ήταν εκτός. Γι' αυτό ε, πήγαμε παραπέρα από τις συστάσεις της ομάδας δράσης αυτής του ΩΣΑ γιατί υπάρχει και επιθυμία στην Ευρώπη να είμαστε στην πρωτοπορία της καταπολέμησης του ξεπλήματος ε, χρήματος ε, και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Καμιά φορά να είμαστε και πιο φιλόδοξοι από το διεθνές πλαίσιο. Επίσης προτείναμε να μειωθεί το κατόφλι από το οποίο κατόφλι και πάνω λαμβάνονται ε, κάποια μέτρα. Μιλάμε για αγαθά υψηλής αξίας, ε, τα κοσμήματα παραδείγματο χάνει. Το κατόφλι ήταν 15.000 ε, ευρώ, το κατεβάσαμε στα 7.500 ευρώ, στα οποία πρέπει να ταυτοποιηθεί ο πελάτης, γιατί ήδη σε κάποια κράτη μέλη είναι πολύ χαμηλό το κατόφλι και είναι στα 2-3.000 ευρώ. Οπότε προτείνουμε να ε, το μειώσουμε στο μισό. Και είδαμε επίσης πως ε, υπάρχουν και φορολογικές παραβάσεις οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν ε, ως πρόδρομα δικήματα, δηλαδή αυτά τα οποία μετά οδηγούν σε ξέπλυμα χρήματος και καταλήξαμε σε αυτά τα οποία τιμωρούνται ε, με το ελάχιστο ενός έτους ε, φυλάκιση και φροντίσαμε μέρα να καλύπτω και τα φορολογικά αδικήματα. Μία μεγάλη αλλαγή στο διεθνές πλαίσιο είναι το γεγονός πως ε, οι προδιαγραφές πλέον δίνουν πολύ μεγαλύτερο βάρος σε αυτό το οποίο ονομάζουμε μία προσέγγιση με βάση την αξιολόγηση κινδύνου. Δηλαδή πρέπει να κοιτάμε τους συγκεκριμένους κινδύνους στις επιχειρήσεις, στο τομεακό επίπεδο, στο εθνικό, στο υπερεθνικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, αναλόγως ε, προσαρμόζουμε και τα μέτρα μας. Γι' αυτό πολλές από τις εξαιρεσει που είχαμε ή έχουμε ακόμα ε, προτείνουμε να μην διατηρηθούν αλλά να εργαστούμε με αυτή την προσέγγιση, να γίνεται δηλαδή μια αξιολόγηση κινδύνου και να μπορέσουμε με βάση αυτή να δούμε ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα. Και αυτή είναι μια σοβαρή βελτίωση στο διεθνές επίπεδο που μπορεί να υιοθετηθεί και στην πρότασή μας. ως αντιστάθμισμα, αν θέλετε, της ευελιξίας και άρα της αβεβαιότητας που εισάγεται εδώ πέρα, ζητήσαμε από τις εποπτικές αρχές στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να δώσουν κάποιες κατευθύνσεις όσον αφορά το τι γίνεται με την αξιολόγηση κινδύνου και έχουμε ορίσει κάποιους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση κινδύνου. Και οπωσδήποτε θα απαιτηθεί περισσότερη δουλειά στην οδηγία και στο μέλλον νομίζω πως ε, θα δούμε στο μέλλον αν θα είναι κάπως πιο ανοιχτή ή κλειστή η οδηγία. Αλλά πρώτα απ' όλα θα εξετάσουμε τον κίνδυνο και μετά θα μιλήσουμε για προσαρμογές. Επίσης, έχουμε εργαστεί στον τομέα της ε, πραγματικής ε, ιδιοκτησίας, δηλαδή ποιο είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης ενός νομικού προσώπου, όποια μορφή και αν έχει. Και φτάσαμε στον ορισμό του ότι κάποιος συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία όταν έχει τουλάχιστον 25% μιας εταιρείας και όποιος έχει τουλάχιστον το 25% πρέπει να ταυτοποιείται για να έχουμε ένα πρώτο επίπεδο όχι, μάλλον, όχι μόνο στο πρώτο επίπεδο, αλλά όπως είπα να φτάνουμε μέχρι το φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από, μια, από το ένα νομικό πρόσωπο, ό,τι μορφή και αν έχει. Επίσης, ξέρω πως ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ πέρα, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για το ζήτημα της ε, προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εδώ πέρα βεβαίως πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ διαφορετικών δικαιωμάτων γιατί η καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος αφορά και τις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ε, και μιλάμε για πράγματα τα οποία πράγματι εξαρτώνται από την διαθεσιμότητα και συλλογή δεδομένων αλλά υπάρχουν και πολλές πολλά ουσιαστικά θεμελιώδη δικαιώματα, δηλαδή το τραπεζικό απόρριτο των ε, ανθρώπων. Μετά από προσεκτική σκέψη λοιπόν εντός της Κομισιόν, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως το υφιστάμενο πλαίσιο όπως ε, εφαρμόζεται είναι το κατάλληλο μέσο και έχει τις απαραίτητες δυνατότητες αλλά και δικλείδες ασφαλείας για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του ξεπλήματος χρήματος. Οπότε, τι κάνουμε, μένει το γενικό πλαίσιο ως έχει στον ε, τομέα καταπολέμησης του ξεπλήματος χρήματος. Έχουμε κάποιες διευκρινήσεις ε, που συχνά αποτελούν αντικείμενο διαφόρων αιτιολογικών σκέψεων Συγκεκριμένα ξεκαθαρίσαμε πως η καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος ε, και της τρομοκρατίας αποτελεί ε, σημαντικό στόχο δημοσίου συμφέροντος ε, αλλά βεβαίως τίθεται και το ζήτημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επίσης λέμε πως τα δεδομένα που συλλέγουν διάφορε εταιρείε και ιδιαίτερα οι τράπεζες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους ε, εμπορικού σκοπούς και τέλος θα έχετε ίσως δει πω υπάρχει ένα αρκετά εκτεταμένο κεφάλαιο για τις κυρώσει που ακολουθεί τη γενική προσέγγιση τη Κομισιόν σε όλη την ομοθεσία για χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε και στο πρόσφατο παρελθόν έγιναν αλλαγές ε, σε αυτό το οποίο προτείνουμε στην τέταρτη οδηγία κεφαλαιακής επάρκειας και οπωσδήποτε θα πρέπει να αλλάξουμε την ε, πρότασή μας ε, στον τομέα των κυρώσεων. Αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα είναι το, αυτό το οποίο προτείνουμε γενικώ με κάποιες προσαρμογές βεβαίω για τη συγκεκριμένη οδηγία. Είναι μια γενική προσέγγιση, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο λοιπόν και ε, νομίζω εδώ μπορώ να σταματήσω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Στρέφουμε τώρα προς την εισηγήτρια κυρία Σαρτζεντήρη πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πόσο χρόνο έχω. Απαντάει χωρίς μικρόφωνο η Πρόεδρος. Εντάξει, θα προσπαθήσω πάντως να μην μακρηγορήσω. Θα είμαι σύντομη. Πρώτα απ' όλα, Ας διαβάσουμε τον τίτλο της ε, οδηγίας «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοδοτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας». Και νομίζω ότι είναι ουσιώδος σημασία εδώ στην Επιτροπή ε, Δημόσιων Ελευθεριών να μην λησμονούμε τον πλήρη τίτλο αυτής ε, της οδηγίας υπό το φως και τη συζήτηση που είχαμε και με την Οικονομική Επιτροπή. Εδώ ασχολούμαστε με αδικήματα μεγάλα άλλα αδικήματα, αλλά ασχολούμαστε και με θέματα τρομοκρατίας. Δεν είναι βέβαια δικιά μας αρμοδιότητα όλα αυτά τα θέματα. Αυτό που θεωρώ ουσιαστική σημασία στη συζήτηση είναι να δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ισορροπήσουμε αντικειμενικά αποτελεσματικό, αποτελεσματικό τρόπο ε, καταπολέμησης ε, της ε, νομιμοποίησης της εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όμως σεβόμενη την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα ήθελα να μελετηθεί περισσότερο η πρόταση αυτή που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προσέγγιση βάσει αξιολόγησης κινδύνου. Γιατί εδώ υπάρχουν κάποια προβλήματα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε όλοι ότι πιστεύω ότι πρέπει να βασιζόμαστε σε σωστές πληροφορίες. Πολλά προβλήματα μπορούν να λυθούν όσον αφορά τη διαφάνεια, εάν γνωρίζουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Ε, όχι να ξέρει η κάθε εταιρεία ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης, αλλά να το ξέρει και το κοινό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια για τα θέματα αυτά. Και επομένως ε, θα πρέπει και στα δημόσια καταστατικά να υπάρχει ε, ο πραγματικός φυσικός ιδιοκτήτης, αυτή η beneficial ownership, δηλαδή να είναι σαφής και να ε, δημοσιεύεται. Θα σας δώσω εδώ και κάποια στοιχεία. το ποσό ξεπλήματος χρήματος έφτασε τα 1,63 ευρώ το 2009 και η υπηρεσία, η, υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για την καλαπολέμηση ε, του ε, εγκλήματος ε, λέει ότι αντιπροσωπεύουν τα χρήματα αυτά 3,6 του παγκόσμιου ΑΕΠ και 60 δις ευρώ κάθε χρόνο ε, περνούν μέσα από παράνομες χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, πράγμα που σημαίνει ότι ειδικά σε αυτή την ε, περίοδο κρίσης ε, χάνουμε πόρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί μέσα από την μη καταβολή των φόρων. Υπήρξε πρόσφατα και μία μεγάλη διάσκεψη ε, για την κίνηση των ε, παράνομων ε, χρημάτων, αυτών των χρημάτων που ξεπλένονται δηλαδή. Επίσης, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων έγινε μία ακρόαση σχετικά με τα φορολογικά δικήματα, αλλά βεβαίως πρέπει να ξέρουμε ε, ακριβώς τι εννοούμε στις χώρες, στις διάφορες χώρες, τι εννοούμε με την έννοια φορολογικό αδίκημα και ε, κατά αυτή την έννοια πρέπει οπωσδήποτε να καταπολεμήσουμε οποιαδήποτε μορφή φορολογικού αδικήματος και επομένως η οδηγία αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθεί και με την φοροδιαφυγή γιατί ε, νομίζω ότι κανένας πολιτικός δεν πρέπει να έχει οποιοδήποτε πρόβλημα επιβάλλοντας τη σωστή φορολόγηση για όλους. Θα ήθελα τώρα να δούμε και κάποια άλλα σημεία και μετά θα σταματήσω. Να πω για μία ακόμα φορά ότι ο καλύτερος τρόπος ε, για να ε, ε, έχουμε σωστή πρόληψη και του ξεπλήματος και της χρηματοδότησης της δημοκρατίας είναι να ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Πρέπει να ξέρουμε δηλαδή ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες και ποιοι είναι οι κίνδυνοι και νομίζω ότι εάν υπάρχει δημόσια ε, πρόσβαση στα Μητρώα, τότε θα βελτιωθεί πολύ η κατάσταση υπό το φως της καταστάσεως όπου ε, κάποιες επιχειρήσεις προσπαθούν να πάνε σε διάφορους φορολογικούς παραδείσους, σε μέρη που θα πληρώσουν λιγότερους φόρους, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι οι πληροφορίες ε, για τις ε, επιχειρήσεις αλλά και για τα μεμονωμένα άτομα τα οποία προσπαθούν να ξεπλύνουν ε, τα χρήματα που έχουν στη διάθεσή τους να αφορά και ανθρώπους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ασχολούμαστε λοιπόν με την εξέβρεση τη πραγματική ιδιοκτησία και αυτό ο πραγματικό ιδιοκτήτη, ο beneficial owner, βρίσκεται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό να γίνεται γνωστό. Μία άλλη ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά αυτήν την προσέγγιση βάσει αξιολόγηση κινδύνου. Πώ εμεί, σαν δημοκρατικά εκλεγμένοι πολιτικοί που είμαστε, μπορούμε να ελέγξουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η ανάλυση και να διασφαλίσουμε την ε, δημοκρατική διαδικασία και την ε, προστασία των ε, προσωπικών στοιχείων. Λέτε ότι η υπηρεσία δράσης ε, κατά του χρηματοπιστωτικού εγκλήματος ε, ε, καταχωρίζει αυτές τις πληροφορίες, ναι, αλλά πού και έχουμε πρόσβαση εμείς στις πληροφορίες αυτές. Επίσης, και όσον αφορά τον άλλο φάκελο που μας ενδιαφέρει όσον αφορά ε, τις ε, σχέσεις ε, αυτών των θεμάτων με τα πολιτικά κόμματα, πώς μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Οπωσδήποτε εμείς θα πρέπει να δούμε όλα αυτά τα θέματα υπό το φως των ελευθεριών των πολιτών και οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να δουλεύουμε. Γιατί είναι προβληματικό, κοντεύει να τελειώσει η θητεία μας και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα ε, να ε, ολοκληρώσουμε την νομοθετική διαδικασία για την νομιμοποίηση εισόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ο κύριος Κίρκοπ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καταστήσω πολύ το σαφέ καταρχά ότι είναι πρόφανες ότι τα θέματα αυτά τα δύο είναι κάτι το οποίο είναι κοινό για την Επιτροπή μα. Ακούμε την Επιτροπή, ακούσαμε και τους συναδέλφους και ο στόχος είναι να ασχοληθούμε με μία εγκληματική απειλή πάρα πολύ σοβαρά. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας να παραμείνει υπεύθυνη η αρμόδια Επιτροπή. Εγώ θα ασχοληθώ σαν ε, κάποιος ο οποίος ασχολείται με την τεχνική ε, πλευρά. Η κυρία Σαρτζετίνη θα είναι στη δημοσιότητα και εγώ θα ενεργώ από τα μετόπισθεν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν οι αρχές αποφάσισαν να επιβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι κανονισμοί θα εφαρτωθούν με τρόπο επαχθέστατο για κάποιους μικρούς ε, επενδυτές, τα πράγματα ήταν δύσκολα, διότι υπάρχει δυσαναλογία δυσκολίας και φόρτου εργασίας. Εγώ είμαι, όπως ε, ξέρετε, ε, σκιώδης εισηγητής στο δικό τη των μέρων. Δεν ξέρω αν εκείνη στο δικό μου το μέρο. Καταλαβαίνετε. Ο καθένα λοιπόν κάνει ένα μέρο ενό όλου. Είναι πολύ λοιπόν ιδιόμορφη η σχέση που θα έχουμε για αυτά τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, πολύ σύντομα, επιτρέψτε μου να κάνω μια-δυο παρατηρήσει. Και πάλι θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα. Ό,τι και να κάνουμε πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν κάνουμε κάτι το οποίο γίνεται τόσο επαχθές και τόσο γελία ε, πολύπλοκο για τους μικρούς επενδυτές ή για αυτούς οι οποίοι μεταφέρουν μικρά χρηματικά ποσά. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός και φαντάζομαι ότι εδώ γίνεται ότι μιλούμε για δισεκατομμύρια. Πήρε κάποιες ε, στατιστικές από το βοηθό μου με κάποια δις και ξέρουμε πόσο κοστίζει το οργανωμένο έγκλημα στα κράτη-μέλη και μέρη και στους Ευρωπαίους φορολογούμενους κάθε χρόνο. Η διαφθορά, όπως καταλαβαίνετε, στις κοινωνίες και οικονομίες μας είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι, ένα από, είναι μία πτυχή μόνο, αλλά από τα πιο άσχημα. Ένα κόμμα. Τρία περίπου τρεις και προσπάθησα σήμερα να καταλάβω τι σημαίνει ένα τρει. Ίσως μπορεί να με βοηθήσει η κυρία Σαρτζαρτίνη. Χίλια δισεκατομμύρια. Εντάξει, αν κάνω σωστά τον υπολογισμό, αυτό μας κοστίζει το ξέπλυμα του χρήματο ετησίω. Και βεβαίω, δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυτόνομο αν θέλετε στον κόσμο του εγκλήματος δεδομένου ότι έχει ε, διακλαδώσεις ε, στην ε, λαθρεμπορία όπλων, στην ε, εκμετάλλευση ανθρωπίνων όντων, σε όλους τους άλλους τομείς διακλαδώνεται. Πρόκειται λοιπόν για χρήματα τα οποία κινούνται ή κερδίζονται παράνομα και πολλά από τα χρηματοπιστωτικά κέντρα τα οποία αφορώνται από τέτοιου είδους χρήματα βρίσκονται στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν διάφοροι εμπορικοί εταίροι ανά τον κόσμο που θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν εμπιστοσύνη στην ενέργεια αγορά για να επενδύνουν. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα μέσα και να συνεργαστούμε με τον καλά τρόπο ώστε να αποτρέψουμε τέτοιου είδους οικονομικά εγκλήματα και να τα καταδικάζουμε. Ξέρετε ότι το χρήμα δεν έχει ε, σύνορα, οι εγκληματίες το ίδιο, όταν κινούν χρήματα, οι διάφορους πόρους που χρειάζεται για να τροφοδοτήσουν τις εγκληματικές τους πράξεις. Χρειαζόμαστε καλούς κανονισμούς, διαφανείς κανονισμούς, αξιοπιστία και όπως είπα και προηγουμένως, χρειάζεται να είμαστε απολύτως σαφείς και να μην ε, επιβάλλουμε υπερβολικό άχθος και βάρος σε άτομα τα οποία δεν μπορούν να το φέρουν. Δύο αυτοί λοιπόν φάκελοι, όπως σας είπα, είναι στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους, γιατί ο ένας ασχολείται με το θέμα του ξεπλήματος ε, χρήματος για, την, ε, για εγκληματικές πράξεις, αλλά ο δικός μου τομέας, η μεταφορά χρηματικών ποσών, επίσης είναι κάτι το οποίο να ληφθεί σοβαρά υπόψη, δεδομένου ότι είναι μέρος των προτάσεων, όπως είπα, που θα πρέπει να κάνουμε για να έχουμε τις κατάλληλες πληροφορίες όταν πρόκειται να σταματήσουμε τέτοιου είδους μεταφορές χρηματικών ποσών όταν υπάρχουν απειλές. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με απόλυτη διαφάνεια, να είναι απόλυτα γνωστοί οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται το θέμα λοιπόν θα το εξετάσω πολύ σοβαρά. προσπαθήσω να επιτύχω ένα, μια ισορροπημένη εκθέση και με την κυρία Σαρτζετίνη και στη συνεργασία μαζί της θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εκθέσεις οι οποίες να είναι χρήσιμες λαμβάνοντας υπόψη και την ε, πρόταση της Επιτροπής. Χαίρομαι λοιπόν ότι... Ε, χαίρομαι διότι μου δόθηκε ο φάκης αυτός και ελπίζω να σας ε, αποσαφήνισα πλήρως τι απόψή μου. Ευχαριστώ και να έχετε καλές σχέσει να συνεχίσετε τη συνεργασία, λέει η Πρόεδρος. Αρχίζει τώρα η συζήτηση. Η κυρία Ματιό κάνει την πρώτη παρέμβαση. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρου του ΕΛΚ και κυρίως τον Φρανκ Έγγελ, τον σκιώδη συγητή που δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ. Ζητά συγγνώμη για την παρουσίαση αυτή τη οδηγία κατά του ξεπλήματο χρήματο. Είναι κάτι το το περιμέναμε εμεί εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν διαφορετικέ πρακτικέ για να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα χρήματο, όπω τόνισαν οι διάφορε εκθέσει. και αυτέ οι διαφορέ απλώ ωφελούν περαιτέρω αυτού που διαπράττουν τέτοιου είδου εγκλήματα. Μιλούμε για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο από εγκληματικέ οργανώσει. Το θέμα του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο είναι ένα σφαιρικό πρόγραμμα που αφορά όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε και απαιτεί να έχουμε συμπεφωνημένο τρόπο δράσης. Η πρόταση αυτή της Επιτροπής περιλαμβάνει ε, τον κατάλογο των χωρών στις οποίες τέτοιου είδους δραστηριότητες αναπτύσσονται. Κυρίως η Γερμανία, η Γαλλία και η... Έχουν το πρόβλημα αλλά αυτό, αλλά το ποσοστό του που επηρεάζεται πιο πολύ του ε, ΑΕΠ είναι αυτό των μικρών χωρών, όπω η Κύπρος και άλλες μικρές νότιες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το θέμα του ξεπλήματος οικονομίας να είμαστε α, πάρα πολύ ε, ακέραιοι και να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα. Χαιρετίζω την πρώτη επιτροπή, καθώ καθώς και την επέκταση του ε, πεδίου εφαρμογής γιατί ώρα ήταν να περιλάβουμε και τα τυχερά παιχνίδια σε αυτές τις τεχνικές ξεπλήματο χρήματο. Θα πρέπει να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους κανόνες, όπως λέει και η Κομισιό, και χαιρετίζω τις διάφορες διατάξεις για την απόλυτη ταυτοποίηση των δικαιούχων. Διαρωτώ με, μήπως θα μπορούσαμε να πάμε ακόμη πιο μακριά. Επιβάλλει όσον αφορά την ανάλυση των κινδύνων η Επιτροπή μόνο στους επαγγελματίες που ασχολούνται με τέτοιε οικονομικέ δραστηριότητε χωρί να λάβει υπόψη άλλα άτομα που συνδέονται, όπως συμβολεογράφου, δικηγόρου κτλ. Όσον αφορά την ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων, διαιρωτώ με εάν είναι αρκετά αποτελεσματικέ οι αλλαγέ που προτείνονται και πρακτικού περιεχομένου. Θα έπρεπε ίσω να σκεφτούμε μήπω θα έπρεπε να κάνουμε κενικά μητρώα στα οποία να καταγράφεται το σύνολο των τραπεζικών στοιχείων των. Ε, ε, των λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων που μπορούν να επιφεληθούν από τέτοιε δραστηριότητε. Όσον αφορά τι κυρώσει, επίση, βρίσκω ότι είναι κρίμα που δεν προχωρήσαμε ακόμη περισσότερο σε θέματα ε, φοροαπατών. Όπω αποδείχνει η σημερινή κατάσταση στην ε, Γαλλία και εκεί γίνονται πολλά. Θα έπρεπε να έχουμε λοιπόν μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Λυπούμε εξάλλου διότι η Κομισιό δεν έλαβε υπόψη αυτή την αναθεώρηση για να μπορέσει να μετρήσει τους κινδύνου που ε, υπάρχουν από, την, ε, από τους νέους τρόπους καταβολής χρημάτων, τους νέους τρόπους πληρωμής, ηλεκτρονικής, τα γκάφη και άλλα τέτοια συστήματα. Επίσης, οι εκθέσεις δείχνουν ότι η μαύρες λίστες οι διεθνείς δεν έχουν πάρα πολλά στοιχεία. Στη διεθνή λίστα του Γκάφη έχουμε μόνο το Ιράν και μια άλλη χώρα. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα αυτό. Γιατί να μην, μπορέσουμε, γιατί να μην δημιουργήσουμε και μια ευρωπαϊκή κοινή λίστα. Ελπίζω ότι με την πρώτη επιτροπή και με τις δικές μας εκθέσεις θα μπορέσουμε να κάνουμε μια εκβαθέαν αναθεώρηση του συστήματος και να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα χρήματος. Ευχαριστώ κυρία Μπόσκο. Eh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, είμαι σκιώδη συγγήτρια για τους ε, σοσιαλιστές και για το ενδιαφέρον και για το μη ενδιαφέρον κομμάτι του φακέλου. Συμφωνώ με τον κύριο Κέρκο πως ε, πραγματικά το θέμα αυτό πρέπει να μένει στην Επιτροπή μας και πρέπει να φροντίσουμε γι' αυτό να μην πάει στην ΕΚΟΝ. Έχω κάποιες ερωτήσεις τώρα στο κομμάτι των ορισμών. Γιατί σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κέρκοπ ε, πρέπει να φροντίσουμε πράγματι να μην επιβαρύνουμε πάρα πολύ αυτούς που κάνουν ε, μικροσυναλλαγές και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ε, να γίνει κάτι τη στιγμή που πιάνουμε τους ε, ανθρώπους αυτούς που πάνε να ξεπλύνουν το χρήμα εκεί πέρα. Χρειάζονται οι ορισμοί εκεί πέρα, χρειάζεται μια κάποια εναρμόνιση. Αλλιώς ξεφεύγουν. Και όπως και στο θέμα της ε, κατάχρησης δεσπόζουσας χρήσης αγοράς βλέπω πως τα κράτη-μέλη δεν ε, κάνουν τίποτα. Δηλαδή λένε πως θέλουν να κάνουν πράγματα αλλά δεν το κάνουν. Και πρέπει άρα ε, όπως είπα, αν να κάνουμε κάτι να το κάνουμε σωστά. Τώρα για την καταβλέμηση της τρομοκρατίας. Υπάρχουν εδώ πέρα πολλές διαφορετικές οδηγίες, νομοθεσία γενικώ για την καταπολέμηση τρομοκρατίας. Ακούσαμε και από την ε, Κομισιόν πως ε, θα έχουμε αν θέλετε, μια γενική, έτσι, ένα γενικό πλαίσιο. Αλλά το πρόβλημα βέβαιως ε, που πάντα σκοντάφτουμε είναι η καλή συνεργασία, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη σε όλα αυτά τα μέτρα. Αν υπάρχει κατακαιρματισμός, δεν κάνουμε τίποτα, αλλά θέλω να ακούσω τι έχει να πει και η Κομισιόν. Ναι, προστασία δεδομένων τώρα. Θεωρούν πως η σημερινή οδηγία και οι μελλοντικέ όπως θα αλλάξουν είναι ένα καλό μέσο, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ακόμα το τι μορφή θα έχει και ότι θα λειτουργήσει σωστά ή να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα. Πώς το ξέρετε αυτό. Και τέλος, αυτό το οποίο λέει η Κομισιόν για ανθρώπου οι οποίοι δίνουν πληροφορίες και το πώς πρέπει να προστατευτούν. Χαίρομαι επίση για το ότι όλος ο ε, συμπεριλαμβάνεται και το στοίχημα δηλαδή που χρησιμοποιείται συχνά από όσου ε, ξεπλένουν χρήμα. Αυτά για την ώρα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ. Βλέπω θετικά βέβαια στο περιεχόμενο του υπομνήματος αυτού. Βεβαίως πρέπει να ανακαλύπτουμε όλα τα χρήματα από παράνομες δραστηριότητες και δεν θα ε, επιτρέπεται να διοχετεύεται σε νόμιμες επιχειρήσεις. Ούτε δε από νόμιμες ούτε από παράνομες επιχειρήσεις πρέπει να χρηματοδοτείται η τρομοκρατία. Το θέμα είναι λοιπόν πόσο σταματάμε. Όπως Ε, λέει λοιπόν και το ανέκδοτο σε κάποιον που, ε, για κάποιον που ζητούσε οδηγίες η σωστή απάντηση είναι εγώ δεν θα ξεκινούσα από εδώ. Και κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχει μια, ένας αρκετά μεγάλος ε, βαθμός ειλικρίνειας, γιατί λένε... Λέτε εδώ πέρα πως το ότι δεν υπάρχουν ε, πλέον εμπόδια, διευκολύνει και τις νόμιμες και τις παρανόμες επιχειρήσεις. Επίσης και η Συμφωνία Σέγγεν και το ενιαίο νόμισμα βεβαίως έχουν καταστήσει το ξέβλημα των χρημάτων και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τις άλλες εγκληματικές δραστηριότητες πάρα πολύ ευκολότερα. Η συνοριακή έλεγχη λοιπόν δεν χρειάζεται ε, να πάμε σε εποχή πρόσεγγεν, ούτε είναι ανάγκη να σταματάμε κάθε νόμισμα. Αλλά η δυνατότητα συνοριακών ελέγχων ε, θα λειτουργήσει και αποτρεπτικά και θα πιάσει κάποιους. Βεβαίως δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενιαία αγορά ή το ενιαίο νόμισμα για το ξέπλυμα χρήματος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ένα παράξενο συσχετισμό ε, πιθανότατα συμπτωματικός, μεταξύ των ευαίσθητων ε, και πλούσιων περιοχών όπου γίνεται εμπόριο αλλά όχι χρήση ναρκωτικών και κάποιων μαγαζιών που κάνουν ε, delivery φαγητών και ταξιτζίδων και ούτε τα μαγαζιά, ούτε οι πελάτες, ε, ούτε τα ταξί έχουν πελάτες, αλλά λειτουργούν και τα δύο με μετρητά. Μάλιστα. Ξαναπερνάμε τώρα στους ηγητές. Κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορώ να είμαι πολύ σύντομη σχετικά με την ερώτηση του κύριου ε, Κίρχοπ ε, σχετικά με το τι ακριβώς σημαίνουν αυτά τα τρεις και εμένα με απασχόλησε λίγο το ζήτημα. Είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο να συλλάβει κανείς αυτά τα ποσά. Άκουσα την κυρία Ματιέ και την κυρία Μπόσκουρτ και τον κύριο Μπρόνς ε, και τον κύριο Κίρκο βέβαια. Ε, βλέπω ότι υπάρχει πολύ καλή θέληση έτσι ώστε να καταφέρουμε να καταλήξουμε ε, σε κάποια σωστή νομοθεσία. Η κυρία Ματιέ λέει ότι θα πρέπει η προσέγγιση του θέματος όσον αφορά την φοροδιαφυγή ε, θα πρέπει να είναι ακόμα πιο έντονη και ε, ενστερνίζομαι την άποψή της. Άκουσα λοιπόν τα σχόλια, βλέπω το τι έχουμε μπροστά μας να κάνουμε ε, και σας ε, ενθαρρύνω να μου κάνετε συγκεκριμένες προτάσεις ε, με τις συγκεκριμένες σας ιδέες έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, να κάνουμε κάτι σωστό σε συνέργεια με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Επομένως να συγκεντρωθούμε και να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κύρκοπ. Νομίζω ότι αυτή η τελευταία πρόταση της κυρίας Αργεντίνη είναι πάρα πολύ καλή. Πιστεύω ότι έχοντας ακούσει και τα σχόλια των συναδέλφων, ε, ε, ε, όλοι είχαν πολύ θετική αντιμετώπιση και βλέποντας και το τι έχουμε κάνει με το ξέπλυμα του χρήματος μέχρι τώρα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ενώ τελικά καταλήξαμε σε κάποιες ε, ε, σωστές προτάσεις σε υπογενικούς όρους, συχνά τα κράτη-μέλη ερμήνευσαν ε, τις προτάσεις με διαφορετικό τρόπο. Μερικές φορές προς ζημία ιδίως των μικρών επιχειρήσεων. Το είδα αυτό με τις αρχές στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά όχι μόνο οι αρχές. Όταν κάνουμε κάποιες ε, γενικές ε, προτάσεις, αυτές εκλαμβάνονται ως ε, πρόταση αλλαγής των διεργασιών ή των δομών από όλες τις οικονομικές αρχές κτλ. Ε, απ' την άλλη πλευρά ε, είναι γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι η δουλειά τους είναι άλλωστε να καταρτίζουν ε, καταλόγους με το ποιος κάνει τι και, ή ας πούμε με νέες υποχρεώσεις αλλά αυτό τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο που ξέρω καλύτερα έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο βάρος για τις μικρές επιχειρήσεις. Ε, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και αυτά τα οποία ε, προτείνουμε, αυτά στα οποία καταλήγουμε ως προτάσεις θα πρέπει να είναι σωστά και να είναι άμεσα συναρτημένα με το τι ακριβώς περιμένουμε να γίνει. Και υπογραμμίζουμε ότι δεν είναι πάντα απαραίτητο οι χώρες μέλη να πάρουν ένα τεράστιο σφυρί και να αρχίσουν να χτυπάνε, ενώ μπορούν να επιτύχουν ίσως και καλύτερα αποτελέσματα ε, με ένα πιο διακριτικό και κομψό τρόπο. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει η ε, ε, ε, υπηρεσίες, ε, η διοίκηση εθνική των κρατών μελών να διαβάζουν προσεκτικά τις προτάσεις και να μην τις χρησιμοποιούν σαν πρόφαση για να μην κάνουν τίποτα. Στρέφομαι προς την Κομισιόν. Θέλετε να πείτε κάτι πριν να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα γιατί... ε, Έγιναν κάποιες ερωτήσεις προς την Κομισιόν ε, όσον αφορά αυτό που μου είπε ο κύριος Κύρκο που είναι γεγονός ότι είναι πιο τεχνικό το ζήτημα και θεωρήσαμε ότι εκφεύγει ε, του, της νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όσον αφορά αυτό το σχόλιο που είπε η κυρία Σαρτζεντίνη ε, σχετικά με την αναφορά των πραγματικών ιδιοκτητών όταν αυτοί βρίσκονται και εκτός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, στο, στην μονάδα αυτή της χρηματοπιστωτικής μονάδας δράσης το λαμβάνουμε υπόψη μας. Εάν μια επιχείρηση θέλει που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θέλει να, να, να έχει συναλλαγή <clears throat> με τράπεζα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπωσδήποτε η τράπεζα θα πρέπει να ζητήσει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα. Ε, ε, υπάρχουν διάφορα στοιχεία της νομοθεσίας και εμείς λέμε ότι η Ευρωπαϊκή ε, ε, επιχείρηση, επιχείρηση δηλαδή που έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει όλες τις ε, πληροφορίες, θα πρέπει να ξέρει εάν και οι αντίστοιχε χώρες έχουν τα ίδια πρότυπα FTF. πώς ε, ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της προστασίας ε, των δεδομένων, αυτό που έθιξε η κυρία Σαρτζεντίνη. Εμείς προσπαθούμε να το δούμε όσο γίνεται πιο ανοιχτά σε σχέση και με τη λογοδοσία, δηλαδή προς τις, προς τις πολιτικές αρχές κτλ. Όταν μιλάμε για εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο, ε, κατά την άποψή μας ε, δεν πρέπει να ε, αναμειγνύονται θέματα προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα συνδέονται με συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πάντως ε, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ε, το γεγονός της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε όλες τις ε, διαδικασίες οι οποίες θα εφαρμόζονται σε πιο χαμηλό επίπεδο και βεβαίω εδώ θα έχουμε και συνεργασία και με τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων. Ακόμα μια ερώτηση από την κυρία Μπουσκούρτ όσον αφορά την καταπολέμηση της τροποκρατίας. Είναι πολλά τα μέτρα που παίρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι πρέπει εδώ να πω ότι εμείς ε, στην ε, προσπάθειά μας να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα ε, ε, το κάνουμε και ε, έτσι ώστε να αποφευθεί η χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν αναφέρονται άμεσα σε χρηματοπιστωτικά ζητήματα, αλλά που αφορούν την τρομοκρατία. Αυτό που χρειάζεται είναι καλή συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλωστε και εδώ ακόμα δίπλα μου κάθονται συνάδελφοι συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έρχονται από άλλε υπηρεσίε. Έχουμε στενή συνεργασία. Κάτι άλλο να πω στον κύριο Κέρκοπ. Βεβαίω συμφωνούμε απολύτω ότι το πλαίσιο αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άσχημα, ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να επιβληθούν ε, περαιτέρω άχθη στις ε, επιχειρήσει. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίω, θα πρέπει να βρεθεί μια καλή ισορροπία έτσι ώστε να γίνει και η δουλειά μα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως, με τα 17 και 18, ανταλλαγή απόψεων ε, σχετικά με την ε, οδηγία για την ε, ασφάλεια στο, στον κυβερνοχώρο. floor for debate. Please. Κύριο Σλάιτερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις αρχές του έτους έβρεξε πολύ σε μια πόλη στη Σουηδία, στον Νόρισκεπ. Πλημμύρισε ένα υπόγειο. Ως αποτέλεσμα αυτού τα τρένα δεν κινήθηκαν για τρεις ημέρες. Έτσι ε, πρέπει να βλέπουμε την, τις κρίσιμες υποδομές και την προστασία τους. Είναι περίεργο το ότι Λίγοι σερβερ σε ένα υπόγειο διέλυσαν το σύρεδρομικό δίκτυο της ε, Νότιας Σουηδίας. Είναι απαράδεκτος αυτός ο σχεδιασμός. Σήμερα μιλάμε για προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους. Ε. Και ε, αυτό είναι άλλο ένα μέτρο που ακολουθεί σειρά άλλων μέτρων και είχαμε βεβαίως ε, και την ανακοίνωση του 2009 και τα συμπεράσματα της Προεδρίας για μια συνεργασία στην προστασία των δεδομένων. Είχαμε την ψηφιακή ατζέντα του 2010 και βήματα προς μια παγκόσμια κυβερνοασφάλεια του 2011. Υπήρχαν λοιπόν αυτά τα μέτρα και στην ε, τωρινή πρόταση οδηγίας έχουμε δύο πτυχές. Ένα μέρος είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι, αν θέλετε, κάποιο είδου στρατιωτική απειλή και σκεμμένες απειλές και μετά έχουμε το άλλο κομμάτι που αφορά εγκληματίες ή χάκερα. Αλλά αυτό το οποίο δεν βλέπω εγώ και είναι πιθανότερο να συμβεί είναι το γιατί δεν προετοιμαζόμαστε για ατυχήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις υποδομές. Θα μιλάμε για κυβερνοασφάλεια. Γιατί μιλάμε για προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά έχουμε και παραδιάσεις επίσης τέτοιες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα λόγω έλλειψης υπηρεσιών. Και μετά η Κομισιόν κατέρτισε ένα ερωτηματολόγιο για το τι βλέπει ο κόσμος ε, ως απειλή και τι θεωρούν ως πρόβλημα. Και επεσήμαναν τις τράπεζες, ε, την ενέργεια και τις μεταφορές. Οπότε η πρόταση αυτή ε, απαιτεί την εισαγωγή ε, κάποιων ομάδων ε, ταχείας αντίδρασης πληροφορικής και λήψη μέτρων για την ασφάλεια των δικτύων. Και γύρω στις 40.000 εταιρείες θα καλύπτονται γιατί θα πρέπει να περάσουν ελέγχους ασφάλειας, να δώσουν ε, να ειδοποιούν τις αρμόδιες εθνικές αρχές για σοβαρά συμβάντα κτλ. Τι σημαίνει αυτό όμως στην πράξη. Είναι ασαφές γιατί πολλές από τις λεπτομέρειες θα αποφασιστούν σε πράξεις κατεξιοδότηση κτλ. Γι' αυτό ανησυχώ λίγο, γιατί όπως είπα υπάρχει αυτή η διπλή αντιμετώπιση. Και το Συμβούλιο πριν από λίγες μέρες υιοθέτησε μια θέση και τονίζει την σημασία της προστασίας των πολιτικών ελευθεριών, προσωπικών δεδομένων κτλ. Αλλά υπάρχει και αυτή η στρατιωτική λογική όπου τα πράγματα θα είναι εμπιστευτικά και απόρριτα για να μην ξέρει το κοινό το τι κάνουμε. Θεωρώ λοιπόν πως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα το ότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι αντοχή των δικτύων πληροφορικής ανεξαρτήτως απειλής το εάν είναι δηλαδή εσκεμμένη ε, από ξένες δυνάμεις, εγκληματίες ή hacker ή εάν είναι κάποιο ατύχημα. Και αυτό το οποίο είδα εγώ, όπως σας είπα, με το περιστατικό στη χώρα μου, είναι πως τα περισσότερα προβλήματα οφείλονταν σε ατυχήματα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει καλύτερη ισορροπία μεταξύ των δύο και να φροντίσουμε οι 40.000 αυτές εταιρείε να ε, όταν ε, θα δημιουργήσουν αυτές τις δομές να φροντίσουμε να προστατεύσουν τα ε, δικαιώματά μας και τα δεδομένα μας. Και να τα κάνουμε τώρα, όχι σε πράξεις κατά για να ξέρουμε τι θέλουμε να επιτύχουμε. Αυτά θα έλεγα. ξέχασα τώρα τίποτα. Α, ναι, κάτι ακόμα. Έχουμε επίσης τα θέματα των τηλεπικοινωνιών και τα λοιπά και τώρα θα διευρυνθεί η αναφορά αυτή των διαφόρων συμβάντων, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη η σύνδεση. Μέχρι το να φτάσουμε στα προληπτικά μέτρα για να μειωθούν τα μελλοντικά συμβάντα. Θέλω να το τονίσω αυτό και επίσης όλες αυτές οι εταιρείες που θα είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν μια τέτοια πορεία πρέπει να έχουν τις απαραίτητες εσωτερικές δομές για να αντιλαμβάνονται την προστασία των προσωπικών δομένων και των πολιτικών ελευθεριών. Αυτό νομίζω πως είναι η συνεισφορά η δική μας. Έχει κολλήσει λίγο η υπόθεση γιατί υπάρχει διαφωνία μεταξύ της ΙΜΚΟ και της ΙΤΡΕ. Από ό,τι φαίνεται η ΙΜΚΟ κέρδισε, η άλλη επιτροπή δεν είναι ικανοποιημένη. Εγώ λέω να γράψω την εκθεσή μου μέχρι να τα βρουν μεταξύ τους. Ευχαριστούμε κύριε Σλίτερ και Με συγχωρείτε για το πώς πρόφερα το όνομά σας. Λοιπόν, η Κομισιόν τώρα θέλει να παρέμβει. Good morning everybody. Καλημέρα σε όλες. Είμαι ο Γιουζέπε Αμπαμόντε υπεύθυνο του τμήματος τη DG Connect της ομάδας που ασχολείται με τις ε, στρατηγικές για την προστασία του κυβέρνου χώρου. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ασχοληθούμε με ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Η οδηγία ισχύει για όλες τις απειλές, τα ατυχήματα και τους κινδύνους που μπορούν να θέσουν σε αμφιβόλο την ακαιρεότητα και την αντίσταση όλων των συστημάτων και δικτύων. Γεγονότα που γίνονται εκ προθέσεως ή τυχαία. Πλημμύρα, ένα σφάλμα στο σύστημα και τέτοιου είδους γεγονότα καλύπτονται από την πρόταση και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στον ορισμό του κινδύνου και του τυχήματος στο άρθρο 3.3.4 3334 που λέει ότι κίνδυνος μπορεί να είναι οποιοδήποτε γεγονός ή συνθήκες που μπορούν να βλάψουν την ασφάλεια. Και είναι κάτι το οποίο το εξηγήσαμε και στο επεξηγηματικό ε, σημείωμα. Δηλαδή όχι μόνο εκ προθέσεως επιθέσεις αλλά και τυχαία γεγονότα καλύπτονται. Αυτό είναι το πρώτο θέμα το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Δεύτερη παρατήρηση. Όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε να κάνουμε με την ανθεκτικότητα των δικτύων και των συστημάτων πληροφοριών ε, και διαδικασίες οι οποίες είναι πάρα πολύ ζωτική σημασίες για το ε, λειτουργία των συστημάτων, για τις υπηρεσίες ε, ε, οι οποίες ε, στα πλαίσια της ε, σημερινής ηλεκτρονικής κοινωνίας είναι αυτές οι οποίες βοηθούν την υποστήριξη των συστημάτων TPE. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να λεβόψει το γεγονός ότι υπάρχουν τεχνικά και οργανωτικά μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να εξασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα και την αντίσταση των δικτύων και συστημάτων δεδομένου ότι όλο περισσότερο είμαστε σε ένα πλαίσιο αύξησης ε, γεγονότων, ατυχημάτων, όχι πάντα εκ προθέσεων. Και στις ε, ε, σημερινές μας κοινωνίες μπορεί τέτοιου είδους γεγονότα να είναι όλο και περισσότερα βαρύνοντα. Γι' αυτό θα πρέπει να καλλιεργήσουμε την κουλτούρα της ετοιμότητας και του τρόπου ταχείας αντίδρασης. Πρώτα απ' όλα ταυτοποιώντας τους κινδύνους τα οποία μπορούν στα συστήματα πληροφορικής να παρουσιάσουν τα δίκτυα και να έχουμε ταχύ τρόπο αντίδρασης και άμβλησης των επιπτώσεων αν συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτός είναι ο στόχος, ένας από τους στόχους τουλάχιστον της οδηγίας. Ο άλλος στόχος και πάλι, και εδώ μιλούμε για μη στρατιωτικές εφαρμογές, είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να συστήσουμε συνεργασίες ε, και συμπεριληπτικές ανά την Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να σας το εξηγήσω κάπως, δεδομένου ότι βρίσκεται στην καρδιά του άλλου προβλήματος και της πρότασής μας. Δηλαδή, να μπορέσουμε τις διάφορες δυνατότητες που υπάρχουν σε επίπεδο μη στρατιωτικό να τη συγκεράσουμε δεδομένου ότι ποικίλουν. Έχουμε περίπου 10 χώρες που έχουν καλές τέτοιου είδους δυνατότητες πρόληψης και ανταπόκρισης, όπως οι σκανδιναβικές χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, που είναι οι προτεργάτες στα συστήματα αυτά και έχουμε κάποιες άλλες χώρες, εάν μπορούμε να τις υποδιαρέσουμε σε τέσσερις ομάδες, αλλά γενικά έχουμε έναν αριθμό χωρών, των οποίων το επίπεδο δυνατότητας αντίδρασης δεν μπορεί ούτε μακράν να συγκριθεί με αυτόν που βρίσκονται στην Βόρεια Ευρώπη. Και ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των διαφορών. Η διαφορά γίνεται σε μικρούς κύκλους. Δηλαδή έχουμε μικρές ομάδες ατόμων που μπορούν να αντιδράσουν σε περίπτωση κινδύνου ή ατυχήματος, αλλά πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για μικρούς κύκλους που αντιδρούν ε, μεταξύ των 17 κρατών μελών. Οι άλλοι μένουν εκτός. Δεδομένου η η συνεργασία βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Τι κάνει λοιπόν η Επιτροπή. Απαιτεί από τα κράτη-μέλη, τα οποία έχουν καθυστέρηση, να κάνουν κάτι για να ανακτήσουν ε, την καθυστέρηση αυτή και να έχουν μέσα στην διάθεσή τους που θα τους επιτρέπουν σε να, φτάσουν σε ένα ελάχιστο επίπεδο ε, θετικής αντίδρασης. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε συνεργασία που να μην αποκλεί κανένα από τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι καλό για τα κράτη που είναι εκτός συστήματος, αλλά καλό και για τις παραδοσιακά καλές χώρες. Διότι όλες οι αλυσίδες ξέρουμε ότι είναι τόσο ισχυρές όσο ο πιο αδύναμος κρίκος τους. Άρα θέλουμε να ενισχύσουμε τους αδύναμους κρίκους της αλυσίδας για να επιτύχουμε αυτή την ε, ε συμπεριληπτική συνεργασία. Σας ευχαριστώ κύριος Μπρόγκ. Κοιτάξτε, στην ε, ηλικία μου το να ανοίγω το κομπιούτερ είναι τόσο δύσκολο όσο το να δένω τα κορδόνια μου. Αλλά είναι συναρπαστικά αυτά που λέει ο εισηγητή, ειδικά το κομμάτι όπου ανέφερε την διακοπή των συγκοινωνιών για τρει μέρε ω αποτέλεσμα μιας πλημμύρα ενός υπογείου. Βεβαίω η πληροφορική έχει βελτιώσει τις επικοινωνίε, τη λήψη αποφάσεων και, και τις ε, δραστηριότητες γενικότερα, αλλά σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν να έχουμε επικοινωνίες χωρίς πληροφορική ως ε, ένα σύστημα ασφαλείας. Ε, να σας πω τι γίνεται να κάνω μια παρομοίηση, παρομοίωση με το αυτοκίνητο. Πριν από 20 χρόνια αν άφηνα τα φώτα αναμένα θα άδειαζε η μπαταρία και θα ζήταγα από κάποιον βεβαίω να μου ξαναβάλει μπρος. Τώρα όμως γίνεται μόνο με μηχανικό αυτή η δουλειά και αυτό το λέμε πρόοδο. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μάθω εάν μπορεί να γίνει κάτι χωρίς ε, πληροφορική. Λοιπόν, το λόγο έχει πάλι ο συγητής. Ναι, άψω αυτό το οποίο είπατε για τα συμβάντα. Εγώ θα ήθελα, όπως είπα, να αυξηθεί και λίγο η αντοχή απέναντι σε ατυχήματα, γιατί θεωρώ πως ε, αυτό μας απειλεί καθημερινά. Βεβαίω σε μια κατάσταση κρίσης ε, θα αλλάξουν οι προτεραιότητες, αλλά η κρίση δεν είναι το φυσιολογικό, δεν είναι ο πόλεμος η καθημερινότητα, οπότε θα ήθελα, όπως είπα, να εστιάσουμε λίγο στα ατυχήματα. Επίσης, οι 40.000 εταιρείε είναι πολλές. Αποκλείονται βεβαίω οι πολύ μικρές αλλά νομίζω πως ε, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε έτσι και τις εταιρείες να ε, αποκτήσουν μια τέτοια λογική. Δηλαδή, οι εταιρείε βασίζονται στο ότι οτιδήποτε έξω από την εταιρεία λειτουργεί. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως ε, πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες ακόμα και αν δεν λειτουργούν τα πάντα γύρω του όπω θα έπρεπε. Γιατί θα έλεγα πω όλοι ασφαλίζουν το σπίτι τους, αν μου επιτρέπετε μπορεί να κοστίζει 1% του μισθού τους, αλλά αξίζει τον άμα καεί το σπίτι. Το ίδιο και για την κοινωνία. Εάν ξοδέψουμε μισό της εκατό ε, στην ε, αντοχή των δικτύων θα είμαστε πολύ καλύτερα αν συμβεί κάτι. Και ε, κοιτάξτε, αυτό εξαφανίστηκε όταν τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος. Επί ψυχρού πολέμου όλοι σκέφτονταν τέτοια πράγματα είχαμε αποθέματα τροφίμων, καυσίμων, ε, οπωσδήποτε τα σπατάλη χρημάτων. Και πέρσι η Σουηδία ε, έστειλε για παλιοσίδερα και τις 30 ε, ατμομηχανές που είχε, που είχε σε περίπτωση που δεν θα λειτουργούσε το ηλεκτρικό δίκτυο, τι οποίε χρησιμοποίησαμε πριν από δύο χρόνια μόλις, έτσι γιατί δεν λειτουργούσαν. Δεν λειτουργούσε όντω το ηλεκτρικό δίκτυο. Οπότε αυτά τα πράγματα δηλαδή να προγραμματίζουμε και για όταν θα πάνε τα πράγματα στραβά. Είναι λογικό και νομίζω πω ε, το σημαντικό σε αυτή την πρόταση είναι να κάνουν κάτι ανάλογο και οι εταιρείε. Οπότε δεν έχω πρόβλημα με την πρόταση. Απλά θέλω να δούμε λίγο και τα, τα ατυχήματα όπω είπαμε. Θα συζητήσω λίγο και μετά θα συντάξω τη γνωμοδότηση μου. Δεν ξέρω πότε ακριβώς τι θέλετε, αλλά φαντάζομαι θα μου πείτε. Δεν ξέρουμε ακόμα, λέει η πρόεδρο, δεν έχω τίποτα. Ούτε και η γραμματεία. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Σλούτερ. Περνάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι... Δεν βλέπω τον εισηγητή όμως. Θα περιμένουμε. Ε, Δηλαδή υπάρχει του Τουρκία με την Τσεφτέσον που έχει παρουσία. As the rapporteur... Κοιτάξτε, ψηφίζει σε άλλη επιτροπή ο εισηγητής θα περιμένουμε να τελειώσει η ψηφοφορία εκεί πέρα. Οπότε διακόπτεται η συνεδρίαση και ξεκινάμε στις 10.30.

Colleagues, let's uh, continue. Συνεχίζουμε, συνάδελφοι. Το θέμα μας είναι η πρόταση κανονισμού για την ηλεκτρονική τραστοποίηση και υπηρεσία εμπιστοσύνη για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην, εσωτερική αγορά. Τον ε, Ιούνιο του 2012 παρουσίασε η Επιτροπή την Επιτροπή της με στόχο να μπορέσει να δημιουργήσει σε ε, πανευρωπαϊκό επίπεδο εμπιστοσύνη για τα θέματα αυτά των ε, υπηρεσιών ε, ηλεκτρονικών συναλλαγών και κυρίως για να διασφαλιστεί αυτά τα θέματα εμπιστοσύνης διασυνοριακά για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση επιβεβαίωση, υπογραφή κτλ. στα πλαίσια του εσωτερική αγοράς. Ο εισηγητήριος ο κύριος, ο κύριος Ροντ θα κάνουμε ανταλλαγή, πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Όπως ε, ξέρουμε, αυτό το οποίο προβλέπεται είναι η παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης 30 Μαΐου, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 6 Ιουνίου και ψηφοφορία στην συνεδρίαση της 8ης και 9ης Ιουλίου. Ο κύριος Ρόντε, ευχαριστώ πρόεδρε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά ψηφίζαμε στην Επιτροπή Ήτρε και έπρεπε να είμαι παρόν. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να χαιρετήσω την πρόταση Επιτροπής για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπηρεσίε εμπιστοσύνη για ηλεκτρονικέ συναλλαγέ στην εσωτερική αγορά. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω για την για την ε, εκτεταμένη δουλειά που έκανε για αυτή την ε, ε, τεχνικό κανονισμό η Επιτροπή. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, όχι μόνο για να υπάρχει ε, μεταξύ όλων των κρατών μελών εμπιστοσύνη, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι πρόκειται για υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται με ασφάλεια. Είναι λοιπόν πρωταρχική σημασίας να εξασφαλίσουμε το ότι αυτό δεν θα μας κάνει πιο ευάλωτους σε ηλεκτρονικά εγκλήματα, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ε, διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων. Θέλει αυτή η Επιτροπή να κάνει ε, την, ε, δύο οδηγίες ε, σε μία για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Έκανε πολύ σωστά τη δουλειά της Επιτροπή, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια αμφισημίες, κάποια έλλειψη ε, ε, διευκρινήσεων σε κάποια σημεία κατά την ε, άποψή μας η χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε κάποιες χώρες δεν έχει γίνει ακόμη υποδεκτή, πρέπει να γίνει. Είναι λοιπόν σημαντικό να ευρεθεί μια λύση ώστε να μπορέσει να υπάρχει ε, διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπαρχόντων συστημάτων σε ηλεκτρονικό επίπεδο. Και αυτό θα γίνει εάν γίνει ε, σταδιακά βελτίωση και ε, ανάπτυξη αυτού του είδους της υπηρεσίας. Επίσης πρέπει να πω ότι πρέπει ε, τα θέματα ε, ασφαλείας κατά την ε, άποψη μου να γίνουν περαιτέρω σαφή, να υπάρχουν διευκρινήσεις θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε ο κανονισμός, να βάλουμε τον κανονισμό να λειτουργήσει, βλέποντας και την νομική πτυχή του προβλήματος. Εκτός λοιπόν από τα επίπεδα ασφαλείας τα οποία πρέπει να οριστούν, πιστεύω ότι θα πρέπει σε θέματα ε, μηχανισμών ελέγχου αξιοπιστίας ε, ελαχιστοποίησης των κινδύνων ε, προστασίας από κινδύνους να δούμε πώς θα προκαιρεσικήσουμε το θέμα αυτό. Υπάρχουν κάποια άλλα θέματα επίσης με τα οποία θα ασχοληθούν οι συνάδελφοι στην Ήτρε και εγώ θα ασχοληθώ μόνο με το θέμα το οποίο με αφορά. Θα δώσω το λόγο τώρα μέσω στην Κομισιό, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε για την εισαγωγή στο θέμα που κάνατε. Η Επιτροπή συνειδητοποιεί πως σημαντικά είναι τα θέματα που θέσατε. Είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε συζήτηση για τα θέματα αυτά. Όσον αφορά τα επίπεδα ασφαλείας, όπως είπατε, προβλέπουμε ότι αυτό θα αποτελέσει μέρος των ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων, αλλά υπάρχει η δυνατότητα και είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση μαζί σας. Εάν δεν θα πρέπει στην πρόταση να συμπεριλάβουμε και αυτό το θέμα του υψηλού επίπεδου ασφαλείας. Για ληστοχυπή των δεδομένων και προστασία των δεδομένων συμφωνούμε απόλυτα ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποια κριτήρια είμαστε της άποψης ότι η οδηγία για την προστασία των δεδομένων εφαρμόζεται πλήρως και μεταφέρθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη, άρα από νομικής πλευράς και συντακτικής δεν βλέπουμε για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνει εδώ αναφορά στο νομικό κείμενο στις, στα νομοθετικές, αυτές πράξεις. Μόλις εφόσον εφαρμόζεται αυτός ο κανονισμός, όλες οι διατάξεις θα εφαρμοστούν και στον τομέα της ταυτοποίησης. Η πρόταση βασίζεται στην νομική βάση που αφορά την ενιαία εσωτερική αγορά, άρα δεν βλέπουμε να είναι αναγκαίο και να υπάρχει η δυνατότητα να θέσουμε ε, ειδικές, να προβλέψουμε ειδικέ απαιτήσει την προσία των δεδομένων και την ταυτοποίηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άμπραχτ πρώτα απ' όλα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Σρόντε για την ε, εισαγωγή που έκανε και την ε, Κομισιόν για την παρέμβασή της. Νομίζω ότι Συμφωνούμε όλοι ότι η πρόταση αυτή είναι η σωστή πρόταση για να έχουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση στον τομέα αυτό και θα ήθελα να κάνω και κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Η μία φορά τις δικές σας παρατηρήσεις να αφορά τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Θα ήθελα τις ασάφειες να τις αποφύγουμε. Δηλαδή, να κάνουμε κάποιες, να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις, να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις. Αυτό είναι καλύτερο όσον αφορά την εφαρμογή κάποιων όλων των οδηγιών και των κανονισμών. Διότι αν υπάρχουν επικαλύψεις πολλές φορές δημιουργούνται ερωτηματικά. Όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσει, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια βελτίωση και να διευκρινίσουμε περισσότερο τους κανόνες που ισχύουν. Δεδομένου ότι οι κανόνες που ισχύουν σε κάθε χώρα είναι διαφορετικοί και εμείς θέλουμε με τον κανονισμό αυτό να επιτύχουμε περαιτέρω εναρμόνιση. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες και να πω ότι για μένα δεν είναι απόλυτα σαφές γιατί υπάρχουν τόσο διαφορετικοί νόμοι και κανόνες που ισχύουν για την ε, ηλεκτρονική υπογραφή και την ταυτοποίηση. Διερωτώ με λοιπόν. Ο κύριος Μασέντιο Λαβάρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Κομισιόν έκανε πολύ θετικά, ανέφερε πολύ θετικά στοιχεία στην πρότασή της. Η αμοιβαία αναγνώριση και ταυτοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και για την ε, ηλεκτρονική ατζέντα και για την αμοιβαία αναγνώριση στην Ευρώπη. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η προστασία των δεδομένων διασφαλίζεται. Όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται σε, ε, στο εδάφιο 7, ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, όλα τα στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στην προστασία των δεδομένων. Κυρίως όταν αναφερόμαστε σε εγκληματικές ενέργειες, όπως αναφέρει και το άρθρο 2 της πρότασης και στα πλαίσια των προνοιών ε, για τις ε, ηλεκτρονικές υπηρεσίες ε, και για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα στοιχεία να είναι σαφή στην οδηγία. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να καλυφθούν όλες οι πιθανότητες κινδύνου ηλεκτρονικά ε, ε, προγράμματα ασφάλειας, ηλεκτρονική υπογραφή κλπ. Ε, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής γιατί οποιαδήποτε παραβίαση αυτών μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε, ό σε όλους. Οι ανεξάρτητες αρχές βεβαίως οι οποίες θα υποπτεύουν τη διαδικασία θα πρέπει να είναι σε θέση ε, να ελέγχουν ε, όλες τις ε, διαδικασίες. Επίσης, στο παράρτημα θα πρέπει να αναφέρονται και ιδιαίτερα ευαίσθητες περιπτώσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει ο εισηγητής να συναντηθεί με τους σκιώδεις πριν αναφερθεί εν τέλει στην τελική μορφή στα θέματα αυτά. Ο κύριος Ρόνταρτ, ευχαριστώ για τα σχόλια. Νομίζω ότι οι δύο λέξεις είναι οι πιο σημαντικές, διευκρινήσεις και τεχνικές βελτιώσεις. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και βεβαίως θα προσπαθήσω να οργανώσω μια συνάντηση των σκιωδών, έστω και αν αυτό τούτη τη στιγμή είναι δύσκολο, καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω λοιπόν. Επομένως, διευκρίνηση και ε, τεχνική βελτίωση. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε από αυτού και όλοι ε, μπορούμε να πούμε στην Κομισιόν ότι έχουμε εδώ μια καλή πρόταση και όταν θα γίνουν και οι, τεχνικές, και οι διευκρινήσεις και οι τεχνικές βελτιώσεις, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε και τις τελικές μας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Ρόντο. Πολύ ωραία. Πάλι όμως αντιμετωπίζουμε δυσκολία. Γιατί στις 11 και 15 προβλέπεται ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο ε, Warright και τον κύριο Φανχόβερ όσον αφορά τον συντονισμό κατά της θερμοκρατίας. Δεν είναι εδώ αυτοί οι άνθρωποι όμως. Πρέπει να περιμένουμε, πρέπει να τους περιμένουμε. Τούτο σημαίνει ότι θα κάνουμε ένα ακόμα διαλυματάκι για καφέ και θα συνεχίσουμε στις 11 και 4. Uh, λοιπόν, ξαναρχίζουμε μετά το διάλειμμά μας. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη και μάλιστα το τελευταίο για σήμερα είναι μια κοινή συζήτηση με τον ε, κύριο Wainwright και με τον κύριο Ζούλτερ Κρόβερ για, ε, για την τρομοκρατία. Καλωσορίζω λοιπόν τον Διευθυντή της Europol και τον Συντονιστή της Αντιδρομοκρατικής Δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, νομίζω ότι καλό θα ήταν να δώσουμε πρώτα το λόγο στους δύο καλεσμένους μας, πρώτα στον κύριο Wayne Wright, Διευθυντή της Europol, έτσι ώστε να παρουσιάσει στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ την κατάσταση της τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την αναφορά των τάσεων. Μετά προτείνω να ακούσουμε και τον κύριο Σιλντε Κερχόβε, και αφού ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους ε, οι δύο ομιλητές ε, θα ξεκινήσουμε την συζήτηση. Κύριε Γουέιν Ράιτ, μπορούμε να ξεκινήσουμε αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της Επιτροπής. Ζητώ συγγνώμη γιατί έφτασα λίγο καθυστερημένος λόγω κίνησης. Με χαρά σας παρουσιάζω σήμερα την ε, αναφορά τάσεων για το 2013 όσον αφορά ε, τις απειλές ε, τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημοσιεύτηκε σήμερα και θα σας την παρουσιάσω εδώ την έκθεση αυτή. Βεβαίω η δημοσίευση αυτή της ε, έκθεση λαμβάνει η χώρα μετά τα γεγονότα της Βοστόνης στι ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα που έδειξαν ότι ε, και οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν παρόμοιε απειλέ. Ε, θα πρέπει κανείς λοιπόν να ταυτοποιήσει πρώτα και τους κύριους υπέτειου των συμβάντων στη Βοστόνη, αλλά παρόλα αυτά δείχνει και η έκθεσή μας για το 2013 ότι η παρακολούθηση των τάσεων της τρομοκρατίας ε, δείχνει, λέω, ότι ε, πολλές περιπτώσεις είναι τρομοκρατία η οποία αναπτύσσεται ε, μέσα στις ίδιες τις χώρες. και βεβαίως σε περίπτωση οποιασδήποτε, οποτεδήποτε προκύπτει διεθνή διασύνδεση ε, μπορεί να υπάρξει και η συνδρομή του FBI. Το 2013 είχαμε δύο ε, μεγάλες περιπτώσεις τρομοκρατίας, μία στο Μπέκερπορτ στην ε, Βουλγαρία, καθώς επίσης και την περίπτωση που θα θυμάστε φαντάζομαι, μίας, ενός μεμονωμένου τρομοκράτη. 17 ε, ε, λοιπόν απώλειες ζωής είχαμε από τρομοκρατικές επιθέσεις ε, το 12 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση των ε, συλλήψεων σε σχέση με την ε, τρομοκρατία το 2012 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι αντιστρέφεται μια πτωτική τάση που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι το 2012 δηλαδή. Αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι παραμένει ορατός ο, ο τρομοκρατικός κίνδυνος στην Ευρώπη που εκφράζεται και εσωτερικά και εξωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απειλή ε, ξεκινάει, μάλλον κινείται από μια τάση για οργανωμένες δράσεις προς μια νέα τάση για μεμονωμένες ε, δράσεις. Ε, γνωρίζουμε ότι, η τρομοκρατία ε, οθείται από πολλές αρχές μεταξύ των οποίων ε, θρησκευτικά ή ε, εθνικιστικά κίνητρα. Το 2012 διαπιστώσαμε ότι είχαμε αυξημένο αριθμό ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, οι οποίοι ταξιδεύουν προς άλλες χώρες, κυρίως προς τη Συρία, στα πλαίσια ριζοσπαστικών ομάδων. Ε, και βεβαίως ε, στην επιστροφή τους ε, τα άτομα αυτά προφανώς αποτελούν αυξημένο κίνδυνο για τρομοκρατικές επιθέσεις. Στην διαφάνεια αυτή που την βλέπετε και στη, στα έγγραφα που έχετε μπροστά σας είναι ε, ένα συνολικό πίνακας, 219 περιπτώσεις σε 7 χώρες, 26% η αύξηση. Ε, στις περισσότερες ε, περιπτώσεις οι επιθέσεις αυτές έλαβαν χώρα στη Γαλλία και την Ισπανία στα πλαίσια αυτονομιστικών ομάδων. Όπως σας είπα, 17 έχασαν τη ζωή τους, 37 τραυματίστηκαν και την, τον προηγούμενο χρόνο είχαμε και στην Βουλγαρία την ε, έκρηξη ενός ύποπτου πακέτου κοντά στο αεροδρόμιο. Ενδεχομένως ε, η περίπτωση της Βουλγαρίας συνδέεται με την Χεσμολά χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί όμως. 537 συλλήψεις είχαμε ε, και ε, αυτό αποτελεί αύξηση της τάξης του 50% ε, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, κυρίως από την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τις κάτω χώρες μέση ηλικία των συλληφθέντων ακολουθεί πτωτική τάση το 2010 η ηλικία ήταν 32 ετών, τώρα έπεσε την προηγούμενη χρονιά ε, στα 28 έτη και μάλιστα 25 για περιπτώσεις ε, ε, θρησκευτικών κινήτρων στις τρομοκρατικές επιθέσεις. Σύμφωνα τις πληροφορίες που είχαμε από την Eurojust, 149 περιπτώσεις τελεσίδικησαν σε 13 χώρες όσον αφορά ε, τρομοκρατικές ε, ε, επιθέσεις. Σε αυτές τις, σε αυτές τις διαδικασίες 400 άτομα πέρασαν από τη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις 126 ε, τρομοκρατικές επιθέσεις αυτονομιστικού χαρακτήρα είχαμε στην Γαλλία και 46 στην Ισπανία, ενώ 6 ε, επιθέσεις το 2012 ε, είχαν θρησκευτικά κίνητρα. 18 αριστερίστικες οργανώσεις επιτέθηκαν στην Ιταλία, στην Ισπανία και την Ελλάδα. Ε, όμως έχει πτωτική τάση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Όσον αφορά τις συλλήψεις, ε, οι περισσότερες συλλήψεις αφορούν αυτονομιστικά κινήματα. 276 συλλήψεις, περίπου το μισό των, συνολικών συλλήψεων. Είναι ένας αριθμός ο οποίος παραμένει σταθερό στα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά τις συλλήψεις θρησκευτικού χαρακτήρα, ε, αυτές παρουσίασαν μεγάλη αύξηση. Το 2012 είχαμε 159 σε σχέση με 122 σε, σε άλλα χρόνια. Ε, μάλιστα στη Γαλλία ο αριθμός αυξήθηκε, διπλασιάστηκε από 46 σε 91 συλλήψεις. Αριστερίστικες οργανώσεις και αναρχικές. Εδώ έχουμε πτωτική τάση. 24 συλληφθέντες σε 4 ε, κράτη-μέλη τον τελευταίο χρόνο. μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία βλέπουμε κάποιες κοινέ τάσεις. Πρώτον όσον αφορά τη χρηματοδότηση ε, της ε, τρομοκρατίας ε, βλέπουμε και έχουμε μαρτυρίες ας πούμε κοινωνικών χρήσης μάλλον πιστοτικών καρτών, κλοπές κτλ. Υπάρχει και δράση εκτός των ε, συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό ε, εξεκολουθεί να είναι ένας από τους κύριους τρόπους για την συλλογή χρημάτων. Επίσης, χορηγίες ή φιλανθρωπικές δωρεές παραμένουν ένα σημαντικό τμήμα ε, των χρημάτων ε, που χρησιμοποιούνται για την ε, εκπαίδευση των τρομοκρατών καθώς επίσης και εκβιασμούς στα πλαίσια των, δικών, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πολίτες ή μη της Ευρωπαϊκής χώρες, της χώρας. Είχαμε μείωση των ε, των ε, εκρηκτικών μηχανισμών ε, λόγω μεγαλύτερου ελέγχου σε αεροδρόμια κτλ. Είχαμε όμως αύξηση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε πολλές περιπτώσεις πέρσι είχαμε ας πούμε ε, κάποιες επιθέσεις ε, στην Πολωνία και στην ε, Ισπανία οι οποίες απεφεύχθησαν και οι οποίες περιείχαν πολύ σημαντικό αριθμό εκρηκτικών αυτοσχέδιων υλών και πρόδρομων ουσιών. Επίσης, ε, όσον αφορά τα, τις ετάσεις επικοινωνίας, μπορούμε να πούμε τώρα ότι ε, και για την τρομοκρατία και για ε, τις ακραίες βίες οργανώσεις υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει μια κοινή πλατφόρμα επικοινωνίας που δίνει τη δυνατότητα σε τρομοκρατικές οργανώσεις να έρχονται σε επαφή με τους συμπαθούντες βεβαίως. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί μια νέα δυνατότητα δυνατότητα ε, έτσι ώστε και να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους αλλά και να προσιλητίζουν ενδεχομένως νέα ε, μέλη. Επίσης ε, είχαμε επιθέσεις hacker, κυρίως ως υπήρχε η περίπτωση της, των hacker του θρησκευτικού φόρουμ, καθώς επίσης και η χρήση βίντεο για την διάδοση των ιδεών τους. Ε, οι τρεις επιθέσεις του Μοχάμετ Μερά στην ε, Τουλούζη βεβαίως ε, έδωσαν και μία νέα διάσταση σε αυτήν την νέα μορφή απειλή του μεμονωμένου δράστη. Ε, βλέπουμε και περιπτώσεις μεμονωμένων δραστών που έχουν λάβει εκπαίδευση στο Πακιστάν ή στο Αφγανιστάν. Επίσης, να σας πω ότι υπήρξαν συλλήψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ατόμων ε, που ανέπτυξαν την τρομοκρατική τους δράση μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχοντας πάρει εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά αυτήν την έννοια γίνονται προσπάθειες καταστολής. Πάντως, τον Οκτώβριο ε, ε, ε, είδαμε μία περίπτωση επίθεσης με χειροβομβίδα σε ένα παντοπολείο κοσέρ στο Παρίσι της Γαλλίας και ξέρουμε ότι η επίθεση έγινε από άτομα τα οποία προσιλητίστηκαν μέσω του διαδικτύου. Επίσης η Τζιχάντ έχει περάσει από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν και σε άλλες περιοχές. Παρόλα αυτά ε, παραμένουν περιοχές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την τρομοκρατία. Το 2012 η Συρία αποτέλεσε ε, ένα νέο πεδίο ε, προσφυλές για τους τρομοκράτες και η επιστροφή αυτών των ανθρώπων από την Συρία ε, μπορεί να σημάνει αύξηση του κινδύνου. Στην Σουηδία ε, είχαμε ε, συλλήψεις ατόμων που ήθελαν να ταξιδέψουν στην Συρία. Ε, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν άτομα στην, στον ένοπλο αγώνα της Συρίας, άτομα τα οποία θα έχουν λάβει εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως από τις πληροφορίες που έχει η Europol δεν υπάρχει πρόβλεψη για επιθέσεις σε στόχους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τρομοκρατικές ομάδες παραμένουν σημαντική απειλή στην Βόρεια Ιρλανδία. Την προηγούμενη χρονιά ε, ε, είχαμε και την δολοφονία ενός σοφρονιστικού ε, υπαλλήλου στην Ιταλία ο ρυθμός των επιθέσεων και των συλλήψεων αυξήθηκε το 2012. Ε, ε, πρόκειται για συλλήψεις ε, από την, τις μελών της ΦΑΗ, του αναρχικού χώρου και ένας ακτιβιστής της, για την πυρηνική ενέργεια δολοφονήθηκε από την ομάδα αυτή η χρήση πυροβόλων όπλων ε, σημαίνει πως αλλάζουν συμπεριφορά καθώς στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν ε, ταχυδρομικές βόμβες και πρόκειται για κλιμάκωση της βίας όπως ε, ορίζεται και στην προκήρυξη με την οποία αναλαμβάνει ευθύνη αυτής της επίθεσης αυτή η ομάδα. Όσον αφορά τον ακροδεξιό εξτρεμισμό όπως του Μπρέιβικ και της οργάνωσης NSU στην Γερμανία, τα κράτη-μέλη έχουν αυξήσει την παρακολούθηση τη χώρου αυτού και είχαμε αύξηση αστυνομικών μέτρων το 2010. Στο αποτέλεσμα αυτό αρκετά φόρουμ στο ίντερνετ ε, απαγορεύτηκαν ή έκλεισαν μεταξύ ε, των οποίων και τα πιο δημοφιλή γερμανόφωνα. Το Νοέμβριο η Ιταλική αστυνομία συνέλαβε 4 άτομα και έψαξε 17 οικίες σε ολόκληρη τη χώρα ε, σε σχέση με ένα Ιταλικό φόρουμ ενός νεοναζιστικού site, καθώς ε, κατηγορήθηκε το site πως διέσπηρε ε, εθνοτικό μίσος. Επίσης, ε, φαίνεται πως πάρα πολλά site κινητοποιούνται σε αυτόν τον τομέα και οδηγούν σε ριζοσπαστικοποίηση και κινητοποίηση υποστηρικτών. Τα τελευταία χρόνια, επίσης, είχαμε ε, ακραίους υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων και οικοτρομοκράτες, αλλά αυτή τη στιγμή προσελκύονται άτομα τα οποία έχουν τάση ε, να χρησιμοποιούν βία. Συνοψίζοντας, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, τι βλέπουμε όσον αφορά τις ε, τάσεις είναι πως η τρομοκρατική απειλή παραμένει ποικιλόμορφη και ισχυρή. Υπάρχει αύξηση της χρήσης ε, πυροβόλων ε, όπλων από πάρα πολλές τρομοκρατικές και ακραίες ομάδες πως η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερα αντίκτυπο στον τομέα τη νομοκρατίας παρά τις προκλήσεις που υπάρχουν και τα μέτρα λιτότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιθέσεις, παραδείγματο χάρη από ακραία και βία στοιχεία, δεν έχουν αυξηθεί ε, σημαντικά από το 2008. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική είναι σημαντική όσον αφορά την ε, τρομοκρατική απειλή. Άτομα τα οποία πηγαίνουν να πολεμήσουν στο Μαλί μπορεί να αποτελέσουν απειλή όταν επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαμε και αυξήσει των απαγωγών στην περιοχή αυτή όπως είπα και ο εμφύλιος της ε, Συρίας προσελκύει ριζοσπαστικοποιημένους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε αύξηση των ατόμων που ταξίδεψαν στη Συρία πέρσι. Ως απάντηση προς όλα αυτά η Europol ε, δραστηριοποιείται και υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στην καταπολέμηση όλων αυτών των μορφών της ε, τρομοκρατίας και βίαιης ε, εξτρεμιστικής δράσης και με επιχειρησιακή στήριξη όπου αυτό είναι δυνατόν και επίσης ίσως πιο σημαντικό απ' όλα η επιχειρησιακή στήριξη των τελευταίων ετών ήταν ε, πάρα πολύ σημαντική στην ε, διερεύνηση της μοβιστικής επίθεσης στη Βουλγαρία. Μας ζήτησαν βοήθεια την επόμενη μέρα και πέρα από την στήριξη υπό μορφή πρόσβασης ε, στην βάση δεδομένων που έχουμε σε δυνατότητες αναλύσεως, δύο στοιχεία ήταν μοναδική, η μοναδική συνεισφορά της Europol. Μπορέσαμε δηλαδή να καθορίσουμε εξετάζοντας τον τόπο του εγκλήματος ε, το ότι υπήρχε μια τηλεκατευθυνόμενη, ένας τηλεκατευθυνόμενος εκρηκτικός μηχανισμός γιατί αρχικά υπέθεταν πως επρόκειτο για βομβιστή αυτοκτονίας και τέλος ε, μπορέσαμε να βρούμε τον εκτυπωτή που χρησιμοποιήθηκε για να τυπωθούν τα πλαστά διπλώματα οδήγησης ε, των ε, υπόπτων χάρη σε μια νέα τεχνολογία που έχουμε για τα πλαστά έγγραφα και μπορέσαμε έτσι να καταλήξουμε στους υπόπτους. Επίσης βεβαίως ε, εξακολουθούμε να έχουμε το την Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Βομβών που αφορά βεβαίως εκρηκτικές τέτοιες ύλες και τεχνικές λεπτομέρειες ε, που χρησιμεύσε στην περίπτωση των Ιταλών αναρχικών. Επίσης εκπαιδεύσαμε τις αρχές ε, στη δίκτυα εκρηκτικών υλών και τέλος ε, πρέπει να πω πως ξεκινήσαμε ένα νέο πρόγραμμα για να δούμε τι γίνεται με τους ριζοσπαστικοποιημένους πολίτες σε που ταξιδεύουν από και προς τη Συρία και άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Wainwright. Θα δώσω αμέσω ε, τον ε, λόγο στον κύριο Ντοκέρχοβε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Να επαναλάβω λίγο πώς βλέπουμε τις τάσεις με βάση αυτή την εξαιρετική έκθεση και μετά αναφέρω και τι συνέπειες έχει αυτό για την ε, πολιτική στο Συμβούλιο. Για τις τάσεις, όπως είπε και ο Ρόμπ, αντιμετωπίζουμε τρομοκρατία που έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια άλλη που δεν έχει σχέση. Και βεβαίως όσον αφορά το πρώτο μέρος έχουμε μια βελτίωση όσον αφορά το κομμάτι των αυτονομιστικών κινημάτων, ΕΤΑ και ήρα. Άκρα δεξιά βεβαίως είχαμε την επίθεση του Μπρέιβικ πριν από ένα έτος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αύξηση ούτε στη, στα αριστερά και άλλα μονοθεματικά ζητήματα επίσης. Τώρα, κάποια άλλα ζητήματα που σχετίζονται. Πρώτα απ' όλα το ΠΚΚ. Είναι μια οργάνωση που εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στην Τουρκία και σημαντικό είναι ότι μπήκαν στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τρομοκρατικών οργανώσεων και είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να διώκουμε τα μέλη του ΠΚΚ στην Ευρώπη γιατί κατά κάποιον τρόπο βοηθάει την ε, διαδικασία στην ε, Τουρκία. Ξέρετε πως ο Τούρκος Πρωθυπουργό ξεκίνησε μια ειρηνευτική διαδικασία με τον Οτσαλάν, τον ηγέτη του ΠΚΚ και αυτό είναι, ε, θα έλεγα πως έτσι στηρίζεται η διαδικασία. Ο Ρόμπαν ανέφερε την έρευνα στον Μπουργκάς, δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο, πιθανή σχέση με τη Χεσμολά που πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά το πώς συμπεριφέρονται στην Ευρώπη, πώς συλλέγουν λεφτά, κάπως σαν το ΠΚΚ που δεν ε, οργανώνουν επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά εκτός. Ε, πλην του Μπουργκάς βεβαίως ε, και όπως αποφασίστηκε στην Κύπρο. από το 2011 βεβαίως έχει πέσει κατά πολύ ο πυρήνας της Αλκάιντα στο Πακιστάν και αυτή τη στιγμή βεβαίως ε, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ποικιλομορφία και πρέπει και εμείς να αντιδράσουμε ανάλογα. Οι τάσεις ε, είναι προς τρεις κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε έναν ε, πολλαπλασιασμό θα έλεγα συνδεδεμένων ή αδελφών οργανώσεων ε, της Αλκάιντα ε, κάτι το οποίο βεβαίως συζητάνε πάρα πολύ ειδικοί. Έχουμε πολλές ομάδες με τοπικά περιφερειακά θέματα που συμφωνούν όμως με την παγκόσμια τσιχά της Αλκάιντα. Έχουμε τα γνωστά στο Ιράκ και στην Αλκάιντα και προσπάθησαν και κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα Ισλαμικό κράτος ε, στο Ιράκ και στη Αλκάιντα στην Ιεμένη που είναι ακόμη πάρα πολύ επικίνδυνη και είναι πάρα πολύ δημιουργική αν θέλετε από πλευράς εκρηκτικών θέλει να δράσει στην Δύση και να προωθήσει ε, τη δράση της στη Δύση. Η Αλκάιντα στο Μαλί επίσης ε, που αποτελεί αντικείμενο της ε, γαλλικής επέμβασης και δείχνει μια τάση αφρικανοποίησης της Αλκάιντα και μια πιο διαρθρωμένη σχέση μεταξύ της Αλκάιντα στο Μαλί και μιας σχετικής ομάδας στο Μαλί, της Αλ Σαμπάμπ στην Σομαλία και του Μπόκο Χαράμ στην Νιγηρία. Θα ακούσατε για την τρομοκρατική επίθεση που σκότωσε πρόσφατα 187 Νιγηριανούς. Μια άλλη ανησυχητική τάση βεβαίως στη ε, Σαχέλ είναι η σχέση μεταξύ τρομοκρατίας και ναρκωτικών. Δεν θα μπω τώρα σε μια ιδεολογική συζήτηση για το εάν η Αλκάιντα στο Μαλή κάνει εμπόριο ναρκωτικών ή όχι, αλλά ε, και τα δύο αυτά επηρεάζουν την ε, χώρα αυτή και εξηγούν γιατί κατέρευσε τόσο γρήγορα το Μαλί. Και βεβαίως υπάρχει και η Αλσαμπάμπ. Αυτή είναι η πρώτη τάση. Η δεύτερη είναι αυτή που ανέφερε ο Ρόμπ. Έχουμε περισσότερους νέους Ευρωπαίους, νέους Ευρωπαίους, αλλά και ανθρώπους που ζουν στη Βόρεια Αφρική και αλλού και πηγαίνουν εκεί όπου υπάρχουν ε, συγκρούσεις, ε, Σομαλία, η Εμένη κτλ. Προσελκύουν κόσμο, αλλά βεβαίως και η Συρία. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία, αλλά αν δείτε τα στοιχεία που μας δίνουν τα κράτη-μέλη. Από την Ευρώπη μιλάμε για εκατοντάδες άτομα και αν ε, το συνδυάσουμε αυτό και με άτομα από τα Βαλκάνια και τη Βόρεια Αφρική μιλάμε για χιλιάδες πλέον. Ε, σημαντικά νούμερα. Δεν είναι όλοι ριζοσπαστικοποιημένοι όταν φεύγουν, αλλά όταν ζήσουν τον πόλεμο, εκπαιδευτούν, θα ριζοσπαστικοποιηθούν ίσως επιτέπου και αν δεν σκοτωθούν εκεί πέρα, όταν επιστρέψουν στην Ευρώπη θα αποτελούν σοβαρή απειλή για την εσωτερική ασφάλεια. Η τρίτη τάση και η φιάλτης των υπηρεσιών ασφαλείας είναι τα μεμονωμένα άτομα ο μονομένος τρομοκράτης που εμπνέεται από το ίντερνετ χωρίς σχέση με κάποιο πυρήνα της Αλκάιντα ή τοπική οργάνωση Αλκάιντα και μιμείται αυτά που βλέπει στα ΜΜΕ. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί παράγοντες που ενισχύουν ή μπορούν να ενισχύσουν αυτή την ε, τάση και μόλις ανέφερα έτσι, τηλεγραφικά κάποια πράγματα ε, και έχουμε ακόμα πάρα πολλά κράτη τα οποία δεν λειτουργούν στον κόσμο και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Και εκεί πέρα θα μπορέσουν να συνταχθούν και να αναπτυχθούν οι τζιχαντιστές. Αυτά τα μέρη αποτελούν καταφύγιο. Είναι αρκετά αυτά τα κράτη. 2014. Ακόμα είναι ερωτηματικό το τι θα σημάνει η απόσυρση από το Πακιστάν για το ίδιο το Αφγανιστάν, για το Πακιστάν και τις διάφορες χώρες Ιστάν, Τατζικιστάν, ε, Ουσμπεκιστάν κτλ. Και μην ξεχνάτε πως ε, το τι είχε συμβεί στην αρχή της ε, Αραβικής Άνοιξης όλοι το θεώρησαν κάτι το θετικό βεβαίως γιατί ε, είχαν περισσότερα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία, λιγότερη διαφθορά κτλ. Αλλά τελικά είχαμε κάποιες συνέπειες. Πρώτον, ε, διαλύθηκαν οι υπηρεσίες ασφαλείας και δεν υπήρξε κάποια αναδιάρθρωση του κλάδου αυτού και κατά κάποιον τρόπο σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο για έναν υποψήφιο τζιχαντιστή να πάει από τα, τα προάστια της Κασαμπλάνκας και να πάει στη Συρία από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια. Και δεύτερον γνωρίζουμε πως η ανάπτυξη της οικονομίας βεβαίως προσφέρει δουλειές και τα αλλά και η ανάπτυξη δημοκρατίας, αλλά όλα αυτά χρειάζονται χρόνο και η... το ότι δεν προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις ε, σημαίνει βεβαίως απογοήτευση, κάτι το οποίο θα εκμεταλλευτούν οι σαλαφιστές. Εάν δείτε δε τον αριθμό ομάδων ε, τέτοιων στο Σαχέλ από το Μαρόκο μέχρι την Ιεμένη ε, είναι η τάση ανισχυτική. Δεν είναι όλες οι ομάδες βίες, αλλά μέλη αυτών των ομάδων των σαλαφιστών είναι βία. Όσον αφορά το σχίσμα ε, σιητών και Σουνητών, δεν θα επεκταθώ, αλλά έχει κάποιον αντίκτυπο γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ πέρα η τρομοκρατία ως ένας άλλος τρόπος ε, αυτής της διαμάχης και πράγματι οι τωρινές οικονομικές συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται πως δεν ε, επηρεάζουν γενικά την ε, τρομοκρατία. Αυτό είναι θετικό και έκτον βεβαίως οι νέες τεχνολογίες, η διαθεσιμότητα πληροφοριών στο διαδίκτυο βιοτεχνολογία, συνθετικά εκρηκτικά, βιο... βιολογικές επιθέσεις κτλ. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τη χάραξη πολιτικής. Η αξιολόγησή μου είναι πως η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκολουθεί να ισχύει και δεν χρειάζεται να αλλάξει. Η πρόκληση είναι να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική με τρόπο σταθερό και ήπιο σε όλους τους πυλώνες ε, προστασία, πρόληψη και αντίδραση και να υπάρχει περισσότερο η σύνδεση μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής πτυχής της απειλής. Ε, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε πρόσφατα δηλαδή να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από την ε, επιθήκη στο Ιν Αμένας και στο Σαχέλ. Φέραμε τους εμπλεκομένους στις Βρυξέλλες, αρμόδιους για την εξωτερική πολιτική και τα ζητήματα δικαιοσύνης και εσωτερικών και είχαμε ενδιαφέρουσε συζητήσεις στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών τη 7 η Μαρτίου ω αποτέλεσμα ενός εγγράφου που συντάξαμε μαζί με την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να δούμε τι μπορεί να γίνει στην περιοχή του Σαχέλ με το να συνδυάσουμε όλα όσα έχουμε στη διάθεσή μας ε, ΚΕΠΑ ε, δικαιοσύνη και εσωτερικών, καταπολέμηση ναρκωτικών, τρομοκρατίας ε, με έναν τρόπο ολοκληρωμένο και να δούμε έτσι τις πιθανές συνέπειες αυτών των γεγονότων στην εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δούμε τα ζητήματα όπως η προστασία των κρίσιμων υποδομών, ε, πρόληψη, το πρόβλημα της ασφάλειας αεροπορίας, ε, ριζοσπαστικοποίηση και απαγωγές για λίτρα. Και τέλος ε, υπάρχει μια πτυχή αυτής της συζήτηση που είναι η πρόκληση των ξένων μαχητών, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα, πώς μπορούμε να σταματήσουμε τους νέους Ευρωπαίους από το να πάνε Συρία και αν δεν το αποτρέψουμε αυτό, να δούμε τι θα γίνει με την επιστροφή τους. Επίσης, ε, εξετάζουμε αυτό το φαινόμενο γιατί είναι δύσκολο φαινόμενο βεβαίω να, να γίνει καταληπτό. Υπάρχουν ε, διαφορετικές περιπτώσεις. Άνθρωποι ρομαντικοί που θέλουν να βοηθήσουν τον ελεύθερο Συριακό στρατό για να ανατρέψει το καστός Άσαντ. Από την άλλη έχουμε ανθρώπους που είναι ήδη ριζοσπαστικοποιημένοι, που τους στέλνουν εκεί πέρα δίκτυα, υποψήφοι τζιχαντιστές και που θέλουν να πολεμήσουν. Προσπαθούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε στη Europol στις υπηρεσίες πληροφοριών, με τη Frontex και με την Κομισιόν. Μετά πρέπει να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο. Ε, δηλαδή να μην αναχωρήσουν καν αυτά τα άτομα και να προσφέρουμε βοήθεια άμα τη αφήξη τους, την επιστροφή τους. Είναι δύσκολο το θέμα αυτό. Τρίτον, να δούμε μια πιο κατασταλτική προσέγγιση την νομοθεσία δηλαδή στην Ευρώπη. Δεν ξέρω εάν ε, και τα 27 κράτη-μέλη έχουν επαρκή νομοθεσία για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Θα θυμάστε πως μετά την επίθεση του Μερά η Γαλλία αποφάσισε να υιοθετήσει νέα νομοθεσία για να καλύψει ε, την εκπαίδευση για τρομοκρατία στο εξωτερικό που δεν ε, κάλυπτε πριν ο νόμος ε, και δεν ξέρω πώς πρέπει να αλλάξουμε την απόφαση πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι πλέον οδηγία για να καλύψει και τέτοιες περιπτώσεις και ήθελα και η Eurojust να κοιτάξει την, ε, το ποινικό σκέλος, πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ποινική διοικητική προσέγγιση η άλλη πτυχή που είναι μια τεράστια πρόκληση είναι το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τους ε, ταξιδιώτες που βεβαίως αφορά και τη χτεσινή σας απόφαση για τα στοιχεία αεροπορικών επιβατών. Βεβαίως δεν είναι δικιά μου η θέση να σχολιάσω την απόφασή σας, αλλά να πω πως ε, είμαστε πεπισμένοι πως ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σύστημα θα προσφέρει προσθέμενη αξία για να μην ε, έχουμε αυτό το φαινόμενο των ξένων μαχητών και να μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε τους νέους οι οποίοι πάνε στο εξωτερικό για εκπαίδευση, γιατί αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτύχουμε κάτι τέτοιο τέλος. Η τελευταία πτυχή είναι το τι πρέπει να γίνει σε σχέση με τις τρίτες χώρες, ειδικά τις χώρες διαμετακόμισης, η Τουρκία και άλλες πρέπει να συνεργαστούμε για να, να δούμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Ντοκερχόφ. Έξι συνάδελφοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Κύριο Κύρκοπ, Ρομέρο Ματιέ, Έντβελτ, Βακεντάιερ και Μπροντ. Αρχίζει λοιπόν ο γύρο ερωτήσεων και μετά θα δώσω το λόγο στου δύο προσκεκλημένους. Ο κύριο Κύρκοπ πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Wainwright και τον κύριο Kirchhoff για τις πληροφορίες που μας έφεραν, που είναι πάρα πολύ σαφείς και μας βοηθούν. Και να συγχαρώ τη Europol για την έκθεσή της, που είναι παράδειγμα του πώς δίδεται ε, εμπεριστατωμένη πληροφόρηση με συνοπτικό τρόπο σε μια εξαιρετική έκθεση και με πολύ ελκυστικό τρόπο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για την έκθεσή σας. Θα ήθελα να κάνω σχόλιο για το PNR ως εισηγητής. Αλλά ακούγοντας τελευταίες σας παρατηρήσεις ε, σήμερα το πρωί, δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο για να δούμε πώς θα προχωρήσει τα πράγματα. Όπως ξέρετε, εγώ είμαι υπέρχομαι της εκθέσεις, αλλά και όλου του ε, θέματος αυτό που αφορά την περιοχή. Νομίζω ούτως ή άλλως ότι πρέπει να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών και κυρίως των ε, ε, εμπιστευτικών. Η ερώτησή μου είναι εξή. Αναφέρατε πολλές φορές, ε, κύριε Wainwright, το θέμα των τρομοκρατών που δημιουργούνται μέσα στις χώρες που ενεργούν. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που αφορά τρομοκράτες που ενεργούν σε κάποιες χώρες και αναπτύσσουν δραστηριότητες στις χώρες που μεγάλωσαν. Μπορεί κάποιος να γεννηθεί σε μια χώρα, να την εγκαταλείψει και όταν έχει στρατολογηθεί σωστά και έχει μάθει πώς να κάνει τρομοκρατικές δραστηριότητες, κάνει. Τώρα, Όλα εξαρτώνται και από την προσωπικότητα και από την κατάρτιση Και αν αυτά δίδονται, παρέχονται και από το χρήμα που παρέχει την αμοιβή, αν παρέχονται από κάποια χρόνια, γίνεται αυτό κάτι τέτοιο στις χώρες μας, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Η κυρία Ρομέρο Λόπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τις πληροφορίες που μας ε, δώσατε και για το πανόραμα του 2012 και για τον τρομα... τρομοκρατία στην Ευρώπη δεν το ότι αυξήθηκε το οργανωμένο έγκλημα. Όπως είπατε έγινε ένα βήμα διαφορετικό. Δηλαδή από δίκτυα τρομοκρατών περάσαμε σε πυρήνες που ενεργούν. Δηλαδή όλο και περισσότερο χρειάζομαι να έχουμε κάτι το οργανωμένο για να μπορέσουμε να αντισταθούμε κατά των τρομοκρατών. Διότι βλέπουμε τώρα ότι είναι πολύ ε, αποτελεσματικός και αυτός ο τρόπος. Δηλαδή, ε, ολιγομελείς ε, ομάδες που οργανώνονται μεταξύ τους χωρίς να χρειάζονται μια μεγάλη δομή. Και αναφέρω το παράδειγμα της Βοστόνης. Πράγμα το οποίο μας κάνει εμάς τους πολίτες πιο ευάλωτους, γιατί μπορεί κανείς να συνεχίσει να παρακολουθεί τα οργανωμένα και μεγάλα δίκτυα τα τρομοκρατικά, αλλά πώς μπορεί πιο εύκολα να αντισταθεί κατά τέτοιων μικρών τρομοκρατικών πυρήνων. Είναι διαφορετικό το θέμα. Και βεβαίως αυτό έχει και να κάνει και με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων, όπως βλέπουμε και στον πόλεμο στο Μαλί, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να κάνει ό,τι έγινε με την τρομοκρατική επίθεση της ε, Μαντρίτη και να συνδέσει αυτό με άλλε εγκρεματικέ ενέργειε. Αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Αλλά η εμπειρία του τελευταίου χρόνου ε, δεν είναι εμπειρία την οποία αποκομίσαμε από τρομοκρατικές δραστηριότητε στην Ευρώπη. Άρα τι είναι καινούριο εδώ. Μία νέα στρατηγική την οποία θα πρέπει να μπορέσουμε να θεσπίσουμε στην Ευρώπη. Διότι είναι προφανές ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών πρέπει να αναπτυχθούν και πώς, πώς μπορεί κανείς να διεισδύσει στο πλαίσια και στο περιβάλλον αυτών που μπορούν να αναπτύξουν τέτοιου είδους ε, νέες τρομο, κρατικές ε, δραστηριότητες. Έχουμε λοιπόν και πάλι τέτοιου είδους ε, ε, καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται από το μίσος που αισθάνονται κάποιοι νέοι, λιγότερο νέοι στις κοινωνίες τους. Και για να μπορέσουν ε, να το ξεπεράσουν γίνονται τρομοκράτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να ε, πολλαπλασιαστεί, να μεγαλώσει. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι για να το κόψουμε όσο περισσότερο έγκαιρα μπορούμε στη ρίζα. Διαφορετικά θα συνεχίσει να επαναλαμβάνεται και να αυξάνεται. Πιστεύω λοιπόν ότι οι αστυνομικές αρχές και οι διοκτικές αρχές και οι αντιτρομοκρατικές θα πρέπει να λάβουν υπόψη πώς μπορεί κανείς να διεισδύσει σε τέτοιου είδους ε, καταστάσεις για να τις προλάβει. Και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε τις νομοθεσίες ώστε τέτοιου είδους ε, εκρήξεις, μίσους να καταστέλλονται και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Ε, una mayor coordinación en los servicios de información de los respectivos estados. Στα διάφορα λοιπόν κράτη-μέλη θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συντονιστούμε με εσά, με τη Europol, με τη Eurojust. Το θέμα είναι πολύ πλοκό και δύσκολο, διότι είναι σε στεγανά όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών παντού. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε διεθνώς, διότι αν δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών προφοριών των διαφόρων κρατών μελών είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε. Και η ενημέρωση για τέτοιου είδους τρομοκρατικές δραστηριότητε και απειλέ είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρόκειται για νέα μορφή τρομοκρατίας ή πάρα πολύ παλιά. Δεν είναι τόσο νέο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό αντιμετωπίζουμε τώρα τελευταία. Επίσης, θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω κάτι για τα δίκτυα στο ίντερνετ. Δεν υπάρχει καμία διεθνής νομοθεσία για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε και να καταδιώξουμε αυτούς τους τρομοκράτες. Πρέπει κάτι να κάνουμε, κάτι να βρούμε για να τους αποτρέψουμε. Τι είδους νομοθεσία θα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση και να διεισδύσουμε στα στεγανά και στα σκοτεινά του ίντερνετ. Και βεβαίως αυτό ισχύει και για τις ε, χώρες οι οποίες ε, είναι ε, στην Βόρεια Αφρική και έχουν αδυναμίες να αντιδράσουν. Και μία τελευταία ενημέρωση παρακαλώ. Σε σχέση με την οδηγία για την οποία αναφέρατε, σε σχέση με την τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία. Γιατί θα ήθελα να ξέρω επακριβώς περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ. Η κυρία Ματιού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρά τον κύριο Ράιτ για την εξαιρετική παρουσίασή του και την εξαιρετική μελέτη που την συνοδεύει ως συνήθως. Έχω διάφορες ερωτήσεις. Μας μιλήσατε για τις πρόδρομες των εκρηκτικών και είπατε ότι έχουν υποχωρήσει σε σχέση με τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Ξέρω ότι υπάρχει ένας νέος κανονισμός που θα ισχύσει ο Σονούπο, που δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικός. Είδαμε ότι διάφορα κράτη-μέλη είχαν ζητήσει εξαιρέσεις και νομίζω ότι θα κάνει να πέσει ο αριθμός των πρόδρομων ουσιών. Μας είπατε όμως ότι το λαθρεμπόριο όπλο να αυξάνεται. Έχουμε να κάνουμε εδώ με συγκοινωνούντα δοχεία, όπως πάντα. Την προηγούμενη Τρίτη, με τη συνδρομή της Europol, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συνδικάτου Οπλοκατασκευαστών κάναμε ένα σεμινάριο για αυτό το θέμα. Θα ήθελα τα κράτη-μέλη και ίσως ο κύριος Ντεκέρκοφ θα μπορούσε να μας βοηθήσει να μπορέσουν να σας δώσουν περισσότερα δεδομένα. Διότι όντως εσείς δεν έχετε πάρα πολλά στατιστικία στην διαθεσή σας, δεν σας παρέχουν τα κράτη-μέλη αρκετά στοιχεία. Είναι πολύ λίγα τα στοιχεία που σας δίδονται από τη Γαλλία. Και θα ήθελα να ξέρω με τι ίδιους όπλα γίνονται οι διάφορες τρομοκρατικές επιθέσεις. Καλά, σνικόφ άλλα όπλα, τέλος πάντων. Έχουμε διαφορετικά παραδείγματα και νομίζω ότι αν έχουμε περισσότερα στοιχεία θα μπορέσουμε να δράσουμε. Το 2015 θα αναθεωρηθεί η οδηγία περί της κατοχής όπλων, αυτοί που νόμιμα μπορούν να κατέχουν όπλα, αθλητές, κυνηγοί και άλλοι θα αφορώνται, αλλά θα πρέπει χωρίς ε, να τους δημιουργήσουμε πρόβλημα αυτό, να τους κάνουμε να συνειδητοποιήσουν κατά ποια πράγματα. Ξέρω ότι μετά ε, φέρθηκε η οδηγία στην γαλλική νομοθεσία και ξέρω ότι οι αθλητές που τα χρησιμοποιούν υποχρεωμένοι να έχουν χρηματοκιβώτιο για να τα ασφαλίζουν το σπίτι τους. Επίσης, θα πρέπει να ξέρουμε αν το λαθρεμπόριο όπλων το οποίο χρησιμοποιούν ή ε, τρομοκράτες προέρχονται από, όπλα τα οποία, οποία κατέχει κάποιος νόμιμα και τα, τα έχουν κλέψει ή πρόκειται για λαθρεμπόριο όπλων και με καλάσνικοφ. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε στοιχεία και τα κράτη-μέλη θα πρέπει αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή τους να σας τα διαβιβάζουν. Υπάρχει έλλειψη σοβαρότητα εκ των κρατών μελών. Επίσης, στη μελέτη αυτή, όπως και στη μελέτη όκτα που μας παρουσιάσατε πριν από λίγο καιρό, ότι υπάρχουν στην τρομοκρατία, Στι τρομοκρατικέ επιθέσει αύξηση της, ε, τρομοκρα... της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο. Είδαμε στη μελέτη όκτα τι γίνεται με την παιδεραστία Φερρυππίν. Και εδώ ε, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ προσωπικά από αυτά τα στοιχεία και βλέπω ότι πρόκειται για κάτι το πάρα πολύ επικίνδυνο. Τι μπορούμε να κάνουμε, υπάρχει απάντηση στο ερώτημα αυτό. Ούτως ή άλλως πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ε, δημιουργεί πρόβλημα στην ε, νεολαία. Η νεολαία η οποία είναι μια ευάλωτη ομάδα την οποία προσεγγίζουν επικίνδυνοι άνθρωποι και την παγιδεύουν και την στρατολογούν. Τι μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε καλύτερη υπαγνήπηση, να έχουμε μαύρη λίστα των επικινδύνων οργανώσεων. Δεν ξέρω εσείς κύριε Wainwright, ο κύριος Κύρχοφ, Μπορεί να μας πει κάτι. Τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει καλύτερα. Κύριε Κύρχοφ, μας μιλήσατε για το ευρωπαϊκό PNR. Όπως και εσείς και εγώ λυπούμε για την εξέλιξη ψηφοφορίας τες, διότι περιμέναμε πολλά από αυτό το θέμα για να έχουμε καλύτερη πρόληψη των κινδύνων. Ξέρουμε ότι 16 κράτη-μέλη είναι έτοιμα να το θέσουν το σύστημα αυτό σε εφαρμογή, αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας μας οδήγησαν για σκοτεινούς λόγους σε απόρριψη. Δεν του καταλάβαμε, διότι η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το πρώτο κατά την απόψή μου. Και ίσως προσωρινά αποτύχαμε. Τι μπορούμε να κάνουμε στο μεταξύ διάστημα. Περιμένουμε απόφαση της Ολομέλειας για να δούμε εάν αντιστραφεί η κατάσταση. Πράγμα το οποίο ελπίζω. Και ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη ούτως ή άλλως θα μπορέσουν να κάνουν κάτι για να προχωρήσουν. Αλλά αν είχαμε επιτύχει την πληροφορία χθε, θα είχαμε κάτι το οποίο θα οδηγούσε σε περισσότερη ασφάλεια του Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ, κυρία Ιντβαλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Βουενράιτ και στον ε, κύριο Ντεκερκόφ. Ε, η ετήσια έκθεση που μας έδωσε ο κύριος Βουενράιτ είναι πολύ σημαντική, όχι τόσο ίσως για τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, αλλά για τις ε, τάσεις ε, όσον αφορά τώρα τον αριθμό των θυμάτων ε, είναι σαφές ότι στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη ο αριθμός των θυμάτων είναι χαμηλότερος από τις άλλα μέρη του κόσμου και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Η συνάδελφος Ματιό είπε ότι λυπάται για μια ψηφοφορία χθεσινή. Εγώ όμως ε, λυπάμαι ότι ήδη πριν από ένα χρόνο περίπου ψήφισε μια έκθεση που ζητούσε διεύρυνση της ε, ε, πολιτικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αλλά κύριε Ντεκερκόφ, ε, με όλο το σεβασμό, όλα τα χρόνια που σας γνωρίζουμε στην θέση που έχετε τώρα και στη θέση που είχατε πριν, κάθε φορά που έρχεστε, μας λέτε χρειαζόμαστε περισσότερη νομοθεσία, περισσότερη νομοθεσία και ξανά ακόμα περισσότερη νομοθεσία. Εγώ θέλω να δω εάν λειτουργεί η υφιστάμενη νομοθεσία, γιατί κάθε μία τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και οι πιο πρόσφατες, ε, καταδεικνύει ένα ε, γεγονός, δηλαδή ότι ήταν ήδη γνωστοί οι δράστες στην αστυνομία ή στις αρχές. Φαίνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση της Βοστόνης ε, ο ε, νεαρός ο οποίος ε, έχασε τη ζωή του νομίζω είναι αυτός που πέθανε που σκοτώθηκε ήταν γνωστός και τον είχε ανακρίνει και το FBI και παρόλο τον αφήσανε να μπει να βγει από τη χώρα να ταξιδέψει όπου ήθελε κτλ. Επομένως γιατί χρειαζόμαστε επιπλέον νομοθεσία. Επίσης θα πρέπει να δούμε, ίσω να συζητήσουμε με τους συναδέλφους από την Νορβηγία, να δούμε πώ εκείνοι αντιμετώπισαν το θέμα της τροποκρατίας, αν δημιουργήσαν νέα νομοθεσία. Όσον αφορά τώρα τους ορισμούς, αυτό παραμένει ε, ε, μπερδεμένο. Ε, κοιτάξτε, εσείς μιλάτε μονάχα για, αναφέρεστε μόνο σε μουσουλμανική τρομοκρατία; ενώ τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι η, μεγαλύτερη, μεγάλη πλειοψηφία είναι των επιθέσεων είναι αυτονομιστικού, εθνικιστικού χαρακτήρα αλλά νομίζω ότι εξακολουθούμε να έχουμε αυτήν την αιμονή με ένα είδος τρομοκρατίας και με εντυπωσίασε και κάτι που είπε ο κύριος Ράιτ ότι ενδεχομένως αυτά τα, ε, τα, τα, μέτρα ε, της ε, λιτότητας δεν οδήγησαν σε ακραία βία αλλά θα μπορούσαν. Να κάνω μια ερώτηση, δεν έχω καμία απάντηση σε αυτό. Υπάρχουν κινήματα τα οποία φαίνεται ότι έχουν εκλεγεί, όπως ας πούμε η Χρυσή Αυγή Ίσως εδώ πηγαίνω σε ευαίσθητα σημεία, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν δέχονται τις δημοκρατικές αρχές, αλλά χρησιμοποιούν βία και θέλουν ε, να ε, καταλύσουν τη δημοκρατία. Ε, η Χρυσή Αυγή δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να την ονομάσει τρομοκρατική, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σαφές ότι αντιτίθεται στις αρχές της δημοκρατίας. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει αυτό να το ξεχωρίσουμε από τους νέους που ενδεχομένως ταξιδεύουν στη Συρία, ας πούμε ή ε, αυτούς που λόγω της ε, απόλυτης φτώχειας ε, και του κοινωνικού αποκλεισμού ενδεχομένως οδηγηθούν σε ε, ε κινήσεις βίας. Έχουμε περιπτώσεις όπου νέοι Ευρωπαίοι είναι οι νέοι Ευρωπαίοι λέτε, ε, οι οποίοι είναι οι δράστες των περισσότερων, όχι εγώ θα έλεγα νέοι άνδρες οι οποίοι είναι δράστες ε, τρομοκρατικών ε, επιθέσεων. Πολύ λίγες είναι οι νέες γυναίκες. Επίσης όσον αφορά το UPNR, νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον δεν υπήρχε κανένας κρυφός λόγος, ήταν πάρα πολύ σαφής οι λόγοι της απόρριψης θα πρέπει να δούμε δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι χώρες ε, σε μεμονωμένη βάση μπορούν να προχωρήσουν με το σύστημα. Υπάρχουν 16 άλλωστε οι οποίες θέλουν να προχωρήσουν. Ευχαριστώ κυρία Μάκιντάιρ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στην Europol για την ε, παρουσίαση που μας έκανε λεπτομερής και συγκεκριμένη. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η παράγραφος που βλέπω εδώ στο έγγραφό σας που αναφέρεται σε αυξημένη χρήση πυροβόλων όπλων και αυτή είναι μια διαπίστωση η οποία αφορά πολλές τρομοκρατικές ε, ε, επιθέσεις. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είχαμε μαζικά πειρά εναντίον ε, αμάχων σε πολλές περιπτώσεις η πρόθεση χρήση ε, των ε, όπλων και των πυρομαχικών ε, είναι μια ευρωπαϊκή τάση, άρα χρειάζεται ευρωπαϊκή αντίδραση. Έχουμε πολλά εργαλεία και τις τεχνολογικές δυνατότητες έτσι ώστε να μπορέσουμε πιο εύκολα να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους τις εγκληματικές ενέργειες και σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και μοιράσματος καλών πρακτικών. Ε, ξέρω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, υπήρξαν πολλές εξελίξεις ε, θετικές όσον αφορά τον έλεγχο των πυροβόλων όπλων και επίσης έχει δημιουργηθεί και μια ειδική βαλιστική μονάδα στα πλαίσια της αστυνομίας. ενδεχομένως ε, έχει ε, ασχοληθεί περισσότερο, ε, συγγνώμη, μία μονάδα βαλιστικής κατασκοπίας και πληροφοριών. Η Interpol νομίζω έχει ασχοληθεί περισσότερο, δεν θα μπορούσε όμως και η Europol να ασχοληθεί με αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Πρόγκ κύριος Γουένραϊτ είπε πως σημαντικός αριθμός τρομοκρατών ή επίδοξων τρομοκρατών συνελήφθησαν ε, ενώ πήγαιναν ή επέστρεφαν από τη Συρία. Παρακολουθείτε μήπως και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, ή θεσμικά όργανα των κρατών μελών που καμιά φορά υπονοούν πως μπορεί να ξεπεράσουν τα όρια από την ανθρωπιστική βοήθεια που είναι βεβαίω θετική στην χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό των τρομοκρατών. Επίσης ο κύριος Wainwright αναφέρθηκε στη δράση κατά των site που υποστηρίζουν την τρομοκρατία ή τη βία. Οπωσδήποτε βεβαίω θετικό αυτό όμως κάνουν διάκριση μεταξύ αυτών των μηνυμάτων και των απλών πολιτικών μηνυμάτων με τα οποία αυτός και οι άλλοι ίσως διαφωνούν. Μπορεί να είναι πολιτικά ή θρησκευτικά, αλλά πάντα πρέπει να γίνεται διάκριση και γίνεται στις ε, ΗΠΑ ε, όσον αφορά στο πλαίσιο της προστασίας ελευθερίας του λόγου ε, μεταξύ απλών δηλώσεων και προτροπών προς την βία. Επίσης αναφερθήκατε σε μεμονωμένους δράστες όπως και ο ένοπλος στο γαλλικό σχολείο και ο Μπρέιβικ πως άνθρωποι χωρίς κάποιες σχέσεις με άλλους, που φαίνεται πως δεν είχαν αυτές οι δύο περιπτώσεις, ε, πως μπορούμε να προλάβουμε τέτοιες περιπτώσεις ε, εκ των προτέρων. Και εγώ επίσης ε, βρήκα ενδιαφέρουσα την χρήση του όρου εγχώριοι τρομοκράτες καθώς δεν χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο για τους Ιρλανδούς ή τους Βάσκους ε, φαίνεται πως απλά υπονοούμε έτσι τους ε, εγχώριους, ε, αλλά όχι θα έλεγα εγχώριες καταγωγής. Θα μείνω σε αυτά. Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και οι δύο μιλητές μας έδωσαν πάρα πολλά και χρήσιμα στοιχεία. Μετά τις συζητήσεις, μετά τις παρουσιάσεις που έγιναν, βλέπουμε ότι έχουν γίνει πολλές ε, συλλήψεις. Τα οικονομικά εγκλήματα είναι αυτά που είναι η μεγαλύτερη επιλογή για μας. Η ερώτησή είναι αν ένας πολίτης με προσεγγίσει και μου πει ε, εάν τα ε, μεταναστευτικά ρεύματα στην Ευρώπη επηρεάζουν ή έχουν σχέση με την ε, ανάπτυξη κάποιων τρομοκρατικών ε, δραστηριοτήτων. Τι λέω. Θα ήθελα να ζητήσω την κατανόηση των διερμηνέων για να καθυστερήσουμε λίγο, δεδομένου ότι άρχισε λίγο αργότερα από ό,τι προβλεπόταν η συζήτηση σήμερα. Αλλά να σας ζητήσω και εσάς να είστε σύντομοι. Ένα πέντε λεπτά ο καθένας, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Ο κύριος Wainwright, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, ερωτήσεις σας θα τις ομαδοποιήσω αναθέματα, δεδομένου ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στην διάθεσή μας. Πρώτα απ' όλα για τους ορισμούς. Σωστά ο κύριος Μπρόγκς και ο κύριος Κύρχο είπε να είμαστε σαφείς. Τι εννοούμε με κάθε έννοια που χρησιμοποιούμε. Και νομίζω ότι αυτό το λαμβάνω υπόψη για να είμαστε προσεκτικοί και συγκεκριμένοι. Τώρα, τι είναι αυτό το οποίο κάνει ακραίους φανατισμούς όλους αυτούς τους ανθρώπους. Στην έκθεση το αναφέρουμε και σήμερα σας είπα επίσης σε ποιο μέτρο προβλήματα και δεν έχεις όπως αυτά στη δεν δημιουργούν προβλήματα και το ίντερνετ επίσης και πώς οι συνθήκες που ισχύουν σε κάθε χώρα, η κοινωνική συνοχή, υψηλή, ψηλή ανεργία κτλ. μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοιου είδους ακραίες καταστάσεις. Ο κύριος Κύρχορ είπε ότι έχει γίνει πιο συγκεχημένη και δύσκολα να προβλεφτεί η απειλή. Και ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι γίνονται ακραίοι και φανατικοί ε, διότι κάτι τους εμπνέει και στο ίντερνετ είναι κάτι το οποίο σήμερα το αντιμετωπίζουμε. Επίσης, είπαμε πώς, πώς θα μπορέσουμε να διαφοροποιήσουμε τις διάφορες μορφές βίας. Πρέπει να δούμε ποιε είναι ο εθνικός ορισμός σε κάθε χώρο. Τα κράτη-μέλη μας έστειλαν κάποια στοιχεία για να δούμε τι εννοούν με την τρομοκρατία, με τα ακραία φαινόμενα κτλ. Αλλά είναι πολύ πλοκό το θέμα. Επίσης ανέφερα το ίντερνετ και αυτό είναι θέρο που ανέφερε η κυρία Ματιού, η κυρία Ρομέρο Λόπες. Το ίντερνετ είναι σημαντικό. Τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε. Εδώ και χρόνια ασχολούμεθα να κάνουμε ένα σχέδιο που λέγεται Check the Web. Πρόκειται για έλεγχο στοιχείων ανοιχτών πηγών, όπως το ονομάζουμε, και προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα πιο ριζοσπαστικά μηνύματα που περνάμε και τα οποία φανατίζουν άλλους. Και η ταυτοποίηση αυτών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι είναι κάτι που θα μας βοηθήσει. Τώρα, τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε έρευνα για αυτά τις ε, απειλές και τις επιθέσεις ε, και τα εγκλήματα στον κυβέρνοχώρο. Ε, η νομοθεσία μπορεί να μας βοηθήσει. Κάτι άλλο το οποίο θέλω να αναφέρω είναι ότι με τη ΣΥΠΑ ε, με το Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο συνεργασίας για τον έλεγχο και την εποπτείο, εποπτεία των μέσων που χρησιμοποιούνται το ίντερνετ για να γίνονται πιο ακραίοι και ριζοσπαστικοί κάποιοι και να ε, επιτίθενται μόνοι τους βία όπως είδαμε πολύ πρόσφατα. πυροβόλα όπλα. Είναι ένα πρόβλημα όλο και περισσότερο που μας απασχολεί και όπως είπε η κυρία Ματιό δεν έχουμε αρκετά στοιχεία από τα κράτη-μέλη και πρέπει να σας πω ότι η δική μας ε, μονάδα ε, αξιολόγησης της ε, ε, απειλή ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Επίσης αναφέρει το θέμα των βέλτιστων πρακτικών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτι που θα συζητήσω με την Μητροπολιτική Αστυνομία. Υπάρχουν ιδέες και προτάσεις, αλλά όπως είπε και η κυρία Ματιέ, ε, υπολογίζουμε πολλά και στις πληροφορίες θα μας παρέχουν τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τα άλλα θέματα, θα ήθελα να αναφέρω κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό που είπε ο κύριος Μπρόγκς. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε κάποια τέτοια γεγονότα από το να συμβούν. Σωστά είπε η κυρία Μίνσβελ, ότι τις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις είναι γνωστά αυτά τα άτομα, ε, αλλά σε άλλες περιπτώσεις όχι. Στην ε, περίπτωση του βούλγαρου τρομοκράτη δεν... Ε, στην περίπτωση την πτήση των Μπουργκάς δεν ξέραμε τι Υπάρχουν στοιχεία τα οποία είχε ε, το FBI που δεν τα ξέρουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν δεν έχουμε τις απαραίτητες μυστικές πληροφορίες ή τις μαρτυρίες, τα στοιχεία που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στο ε, επίπεδο της πρόβλεψης μιας τέτοιας ε, τρομοκρατικής επίθεσης. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να υπάρχει ε, συνεργασία και μελέτη του τι ακριβώς βλέπει ο καθένας στα διάφορα αυτά, ε, στους διάφορους σχετικούς ε, ιστοτόπους του ίντερνετ. Και πολλές φορές υπάρχουν τότε τόσο πολλά αρνητικά σχόλια για κάποια θέματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε ακραίες καταστάσεις. Ευχαριστώ. Κύριος Δοκύρχοφ. Δεν θα ξανανοίξω το θέμα του ορισμού αυτών των τρομοκρατών homegrown. Απλώς θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια κατηγορία ατόμων που δεν έχουν σχέση με την Αλκάιντα, αλλά δεν ενεργούν πάντα μόνοι τους, διότι είναι σε επαφή με άλλους, σαν τον Μεχά, ε, ταξίδευαν, είδαμε ότι είχε ταξιδέψει ο συγκεκριμένος και είχε σχετιστεί με άλλα υποπτάτομα, αλλά πολλοί από αυτούς πραγματικά δεν ε, οδηγούνται σε αυτό που κάνουν από ομάδες. Πολλές φορές έχουμε να κάνουμε και προσαρμογή των ορισμών που κάναμε έχουμε να κάνουμε με οι ομάδες. Κυρία Ρομέρο Λόπες ρώτησε αν χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική. Όπως είπα, μια στρατηγική όχι, αλλά στον τομέα της πρόληψης, της στρατολόγησης πρέπει κάτι να κάνουμε και να ενημερώσουμε την στρατηγική που είχαμε θέση εφαρμογή πριν από 4-5 χρόνια. Και θα πω, δεν είχαμε μεγάλη εμπειρία όταν ε, πριν από 5-6 χρόνια καταρτήσαμε αυτή την στρατηγική μας. Πολλές χώρες έχουν εμπειρία επιτυχιών και αποτυχιών και φαντάζομαι ότι τις επόμενες μήνες μέχρι τον Νοέμβριο θα κάνει μια ανακοίνωση Επιτροπή για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε περαιτέρω τη στρατηγική μας. Για μένα, τη μεγάλη πρόκληση είναι το ίντερνετ για τρία θέματα. Ξέρουμε τι κάνει για τον εποπτεία τη Europol, αλλά δεν επαρκεί δεν έχει αρκετές πληροφορίες και δεν μπορεί κάθε κράτος μέλος χωριστά από τα 27 να κάνει μόνο του την σχετική έρευνα. Νομίζω ότι από κοινού σε επίπεδο Europol γίνονται πολλά πράγματα. Επίσης, ακόμη δεν ξέρουμε πώς να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τον ιδιωτικό ε, τομέα και τους φορείς παροχής υπηρεσιών για να μπορέσουμε ε, να ελέγξουμε και να κατεβάσουμε από το ίντερνετ αυτούς απαράδεκτους ιστότοπους. Αλλά πολλές φορές αν δείτε τι κυκλοφορεί στο ίντερνετ θα εκπλαγείτε. Όπως είπε και ο Ρόμπ, ίσως το πιο σημαντικό θέμα είναι πώς μπορούμε ε, να κάνουμε ε, κάτι εμείς τους αντίποδες για να μπορέσουμε να αντισταθούμε και να πολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Πώς μπορούμε εμείς στις κυβερνήσεις μας να κάνουμε κάτι για να μην ακούγονται μόνο οι ακραίες φωνές αλλά να αμβληνθεί αυτή, αυτός ο φανατισμός. Είναι λοιπόν προτεραιότητα να αυξήσουμε τα κονδύλια που έχουμε για να ενισχύσουμε τις χώρες που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ακραία τρομοκρατικά φαινόμενα. Οι χώρες αυτές πρέπει να ενισχυθούν και να αναπτύξουν περισσότερο τις δυνατότητες που έχουν να αντισταθούν αυτών. Τώρα, θα ήθελα όσον αφορά τα όπλα να σας πω ότι λαμβάνω υπόψη τα ε, στοιχεία που αναφέρετε. Όντως θα ζητήσω από τα κράτη-μέλη να δίδουν περισσότερα στοιχεία στην Ευρωπόλη όσον αφορά τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Εδώ έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερα από ό,τι σε θέματα κυβερνοασφάλειας και χαιρετίζω το γεγονό ότι με την κυρία Άστον η Κομισιό πρότεινε τώρα μία στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια, διότι πιστεύω ότι με το κέντρο και την Europol ε, με τα μέτρα που έχουμε λάβει έχουμε προχωρήσει αρκετά και έχουμε κάνει αρκετά. Αλλά κάποια μέρα το να μπορεί να μπει στο Σκάντα, σε ένα, μια τρομοκρατική ομάδα, σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο, σε ένα, στα άδυτα ενός ε, αεροδρομίου, θα είναι καταστροφικό. Ο κίνδυνος, ε, λοιπόν, επίθεσης ε, μιας Ενό κρίσιμου έργου υποδομή μέσω ίντερνετ δεν είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουμε ούτε σήμερα ούτε αύριο. Έχω αμφιβολίε. Νομίζω θα πρέπει εμεί να προετοιμαστούμε καλύτερα και νομίζω ότι δεν είναι παρκώς προετοιμασμένα για τέτοιου επιδέσεις στα κράτη-μέλη όσον αφορά το PNR. Θα σα πω ότι είναι παράδοξο το ότι εμεί ε, σήμερα σε μία αεροπορική εταιρεία δίδει εκτό Ευρώπη όλα αυτά τα στοιχεία με περισσότερε λεπτομέρειε από ποτέ και τα κράτη-μέλη πιστεύω ότι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το δικό τους PNR, διότι δίδει εγγύσεις ίση όρους, η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια, διότι αν κάνουν κάτι 16 από τους 27 μόνον, έχουμε πρόβλημα. Έφυγε η Σοφή. Και δεν μπορώ να τις απαντήσω. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι το ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο δεν ήταν... Ε, δεν είμαστε εμείς που ζητούσαμε την αξιολόγηση. Εν πάση περιπτώσει ε, πρέπει να σας πω ότι ε, δεν μπορώ εγώ να κάνω τέτοιου είδους αξιολόγηση για την ε, υπηρεσία πληροφοριών, δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μας. Δεν ζητά όλο και περισσότερα, ζητά όλο και καλύτερα. Ε, ενδεχομένως πρέπει να βελτιώσουμε την νομοθεσία, πρέπει να την προσαρμόσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα όπλα, για τα πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά κτλ. Ε, μπορεί να υπάρχει νομοθεσία, αλλά πρέπει να βελτιωθεί και ε, δεν θέλω να, να δημιουργώ διαρκώ νέα επίπεδα ε, νομοθεσία. Κοιτάξτε, επίσης, εγώ δεν είμαι... Ε, δεν έχω αιμονή, όπως είπε η Σοφή, με, το, με την τρομοκρατία την Ισλαμική. Απλώς διαπιστώνω, άλλωστε δεν την ανέφερα με το όνομά της ποτέ. Εγώ λέω απλώς ότι ε, ε, ε, αντιθέτως πιστεύω ότι δεν υπάρχει άμεση γραμμή ανάμεσα στο Ισλάμ και την τρομοκρατία. Είπα επανειλημμένα ότι στρεβλώνεται, είναι hijacked όπως λέμε στα αγγλικά ή ο Ισλαμισμός έτσι ώστε να καταλήξει στην τρομοκρατία. Όσον αφορά τώρα τις μεταναστευτικές ροές, ε, βεβαίως γνωρίζουμε ε, ε, και τις, τις οδούς της μετανάστευσης, γνωρίζουμε τις παραμέτρους, ενδεχομένως κάποια, κάποια ένταξη καλύτερη να, ε, να βελτιώσει την κατάσταση, αλλά από την άλλη πλευρά ξέρουμε ότι στο Βέλγιο ας πούμε έχουμε 7 ανθρώπους οι οποίοι είναι Βέλγοι, οι οποίοι έχουν γεννηθεί στο Βέλγιο, δεν είναι πρώτη γενιά ή δεύτερη γενιά μεταναστών και οι οποίοι όμως ε, τελικά πηγαίνουν στη Συρία γιατί θέλουν ε, να αγωνιστούν σε πλαίσια τρομοκρατικών Ισλαμικών ομάδων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρο. Ευχαριστούμε που ήρθατε και μα είπατε όλα αυτά τα ωραία ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστούμε του διερμηνεί, λέει η Πρόεδρο, που είχαν την καλοσύνη να μα δώσουν περισσότερη ώρα. Oh, uh, good Και ε, καλό μεσημέρι.